Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε παρακαλώ. Καθίστε λοιπόν. Θα ήθελα να σας γνωρίσω τον Μάρκο Μαρινάρη που είναι από τη Γενική Διεύθυνση της Προεδρίας που θα μας παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα λειτουργήσει η Ολομέλεια. Το λόγο λοιπόν στο Μάρκο Μαρινάρη. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι έχετε μπροστά σας μια μεγάλη μέρα 1, 2, 1, 2. Put on your headphones, please. Παρακαλώ, φορέστε τα ακουστικά σας για να έχετε μετάφραση. Γιάννη, εντάξει. Please put on your headphones so that you can hear the Φορέστε τα ακουστικά σας για να ακούσετε ποια θα είναι η διαδικασία, πώς θα δουλέψουμε σήμερα. Αρχίζουμε. Θα σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες. Καλώς ήρθατε πρώτα απ' όλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρίες. Προκειμένου να αρχίσουμε σωστά και καλά, θα δώσω το λόγο στον Μάρκο Μαρινάη από τη Γενική Διεύθυνση της Προεδρίας που θα μας παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ε, διαδικασίες της Ολομέλειας. Μάρκο. Thanks, Pat. Ευχαριστώ Πατ. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι έχετε μπροστά σας μια μακρά ημέρα εργασιών στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο σκεφτήκαμε ακριβώς να ξεκινήσουμε αυτή την ημέρα δίνοντας σας μια σύντομη εικόνα των δραστηριοτήτων αυτού του θεσμικού οργάνου, των μελών του, του τρόπου εργασίας τους κυρίως, διότι σήμερα θα εργαστείτε κι εσείς όπως και αυτοί, όπως εργάζονται αυτοί καθημερινά και όπως εργάζονται στις Ολομέλειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια ιδιαιτερότητα που το διαφοροποιεί από τα άλλα. Γιατί είναι το μόνο θεσμικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες. Όπως σίγουρα γνωρίζετε, κάθε πέντε χρόνια όλοι εμείς καλούμαστε στις κάλπες για να δώσουμε την ψήφο μας. Να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας, οι οποίοι έρχονται εδώ για πέντε χρόνια, ώστε συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους, της Κομισιόν, του Συμβουλίου και των υπολείπων θεσμικών οργάνων τόσο για τη βελτίωση της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας όσο και κυρίως για την εκπόνηση νέων νόμων που πάντα στοχεύουν στη βελτίωση των συνθήκων της καθημερινής μας ζωής. Οι βουλευτές είναι αυτή τη στιγμή 754 και εργάζονται στο πλαίσιο ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών, κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών, αλλά επίσης συνεδριάζουν όλοι μαζί σε αυτή την αίθουσα και σε άλλες αίθουσες, ώστε να μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις. Όταν τώρα οι βουλευτές ε, κάθονται σε μια αίθουσα όπως αυτή, δεν κάθονται όπως εσείς σήμερα, ανεθνική αντιπροσωπεία, χωρίζονται στις επωνομαζόμενες πολιτικές ομάδες. Γιατί, διότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί με ευρωπαϊκό διεθνικό τρόπο, για αυτό το λόγο οι βουλευτές κάθε χώρας καταφτάνουν εδώ και συνεδριάζουν βάσει των πολιτικών τους ιδεολογιών. Φυσικά σήμερα για εσάς η κατάσταση έχει διαφορετικά. Ε, εκπροσωπείτε διάφορες χώρες και φυσικά κάθεστε κατά εθνική αντιπροσωπεία. Όταν οι βουλευτές εργάζονται εδώ σε αυτή την αίθουσα, στις πρώτες σειρές, ε, έχουμε πάντα τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, μαζί με αυτούς οι αντιπρόεδροι, αρχηγοί αντιπροσωπείων, αρχηγοί επιτροπών και πίσω όλοι οι υπολείποι ευρωβουλευτές που κάθονται με αλφαβητική σειρά. Αυτό για να μην δίνεται διαφορετική αξία στους διάφορους βουλευτές. Όταν εργάζονται εδώ οι βουλευτές μπορούν να εκφραστούν στη μητρική τους γλώσσα, όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Και έτσι μπορείτε να πράξετε κι εσείς σε όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Για ποιο λόγο το κοινοβούλιο από την αρχή, από τη δεκαετία του 50, έδινε την ευκαιρία έκφραση στη δική του γλώσσα σε κάθε βουλευτή, διότι εδώ μιλάμε για μια δημοκρατική συνέλευση. Μια συνέλευση όπου κάθε Ευρωπαίος πολίτης είναι εκλέξιμος Συνεπώς, για να μην μπορούν οποιασδήποτε ελλείψεις γνώσης ξένων γλωσσών να αφαιρέσουν από κάποιου ανθρώπου τι ικανότητε να βρεθούν εδώ, ο κάθε βουλευτή μπορεί να μιλάει τη γλώσσα του, τη μητρική του γλώσσα. Και εσεί λοιπόν σήμερα εδώ μπορείτε να μιλήσετε στη δική σα μητρική γλώσσα. Φανταστείτε λίγο μία ημέρα ολομέλειας με παρόντες άνω των 700 βουλευτών και πάρα πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη. Πώς να διαχειριστεί κανείς όλους αυτούς τους ευρωβουλευτές που φυσικά θέλουν να πούν την απόψή τους. Λοιπόν, ε, ορίζονται αυτό που ονομάζουμε χρόνοι ομιλίας. Δηλαδή κάθε πολιτική ομάδα ανάλογα με τον αριθμό βουλευτών που έχει λαμβάνει ένα χρόνο ομιλίας καθημερινά. Όσο πιο μεγάλη είναι μια πολιτική ομάδα φυσικά, όσο πιο πολλά μέλη έχει, φυσικά τόσα περισσότερα λεπτά ομιλίας θα λάβει. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου εκχωρούν το χρόνο ομιλία στις διάφορες ομάδες και μετά κάθε ομάδα αποφασίζει από μόνη της ποιος βουλευτής θα μιλήσει και για πόσο χρόνο. Ο χρόνος ομιλίας ε, κυμαίνεται από ένα ελάχιστο 30 δευτερολέπτων έως το πολύ 6 λεπτά. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές σε μια φυσιολογική ημέρα εργασία όπω η σημερινή λαμβάνει το λόγο για ένα λεπτό, ενάμιση, το πολύ δύο. Ίσως να σας φανεί περίεργο. Θα μπορούσατε να αναρωτηθείτε, μα τι να προλάβει να πει ένα βουλευτή σε ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό. Στην πραγματικότητα καταφέρει να πει πολλά. γιατί, διότι η Ολομέλεια πρέπει να θεωρείτε ότι είναι το σημείο τερματισμού των συζητήσεων που έχουν ήδη λάβει χώρα στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου, στις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο, όταν ένα βουλευτή σηκώνεται για να πάρει το λόγο, παρουσιάζει ουσιαστικά μόνο τα συμπεράσματα της εργασίας του, διότι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές γνωρίζουν ήδη τι έχει κάνει. Έτσι θα εργαστείτε κι εσείς. Φτάνετε εδώ, όπως είναι φυσικό, με σαφείς προτάσεις που αποτελούν ε, ε, αποτέλεσμα των συμπερασμάτων σας. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα λάβετε μια λίστα των ομιλητών. Θα, ο πρόεδρος που διευθύνει τη συνέλευση θα καλεί τον ομιλητή να λάβει το λόγο και θα δείτε ότι στις οθόνες που έχουμε εδώ δεξιά και αριστερά μας θα αρχίσει να τρέχει ο χρόνος. Αυτό δεν είναι απειλή, ε. Είναι απλά για να σας βοηθήσει. Να θυμάστε ότι αν χρειαστεί να μιλήσετε και σας δόθουν δύο λεπτά θα πρέπει να τηρήσετε αυτό το χρόνο. Φυσικά, εάν στο πέρα των δύο λεπτών δεν έχετε ολοκληρώσει την πρότασή σας ή την ομιλία σας, κανένα δεν θα σας διακόψει ξαφνικά. Θα σας δοθούν και κάποια δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε. Αλλά σας παρακαλούμε να μην καταχραστείτε το χρόνο που σας εγχωρείτε. Και αυτό επαναλαμβάνω ώστε να δίνετε η δυνατότητα να μιλήσουν όλοι οι ομιλητές. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ μην θεωρείτε ότι σας θερούμε την ελευθερία λόγου. Θεωρήστε το ως μια ε, σωστή συμπεριφορά προς τους ε, συνομιλητές σας ώστε το πρόγραμμα να μπορέσει να διεξαχθεί σωστά και ομαλά μέχρι το τέλος. Αυτή η αίθουσα στην οποία σας υποδεχόμαστε σήμερα δεν είναι η αίθουσα της Ολομέλειας κανονικά οι εργασίες σας θα λάμβαναν χώρα εκεί. Ωστόσο, η αίθουσα της Ολομέλειας που βρίσκεται στην άλλη πλευρά από τις σκάλες, απέναντι από αυτή την αίθουσα, είναι κλειστή προσωρινά για εργασίες ανακαίνησης. Γι' αυτό τον λόγο αποφασίστηκε να υποδεχθούμε τις εργασίες αυτής της Συνόδου σε αυτήν εδώ την αίθουσα. και να προβλέψουμε και μια αίθουσα ακρόασης ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν σε κάθε περίπτωση να παρακολουθούν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Η ολομελιά σας ε, είναι πολύ πλούσια, περιλαμβάνει πολλά θέματα γιατί συγκεντρώνεται, συμπτύσσεται σε μία μόνο μέρα. Όταν οι βουλευτές συνεδριάζουν σε ολομέλεια, κανονικά συνεδριάζουν για τέσσερις ημέρες αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ημερών είναι αρκετά εντατικέ οι εργασίες. Φανταστείτε ότι ξεκινάει κανείς το πρωί στι 8.30 με 9, εργάζεται μέχρι την ώρα του μεσημεριανού, μετά λαμβάνουν χωρί ψηφοφορίε και μετά από αυτές ε, ξεκινάνε ξανά οι εργασίες γύρω στις 3 μέχρι τις 8, διάλειμμα για βραδινό και μετά από τι 9 μέχρι τι 12 τα μεσάνυχτα. Και αυτό από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Για ποιο λόγο πρέπει να δουλεύει κανείς τόσο εντατικά, διότι μέσα στα χρόνια αυτή εδώ η κοινοβουλευτική συνέλευση κατάφερε να λάβει όλο και περισσότερες εξουσίες. Ακριβώς λοιπόν αυξάνοντας τις εξουσίες της αυξήθηκε και ο φόρτος εργασίας και η νομοθετική φάκελη προσυζήτηση για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν μαζί όλες αυτές οι εργασίες ώστε να διεκπαιρεωθούν όλοι αυτοί οι φάκελοι που επαναλαμβάνουν είναι πολύ άριθμοι, όλο και περισσότεροι και για ποιο λόγο είναι όλο και περισσότεροι. Διότι στην Ευρώπη σήμερα έχουμε ένα σύστημα ε, δύο κοινοβουλίων ουσιαστικά. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβουλίο των Υπουργών που έχουν ίσες εξουσίες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει πολλή δουλειά, πολλή δουλειά διότι τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμιοδιότητες σε σχεδόν όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Σκεφτείτε ότι σήμερα πάνω από το 80% της νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεταφορά ευρωπαϊκών νόμων ουσιαστικά νόμων που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, την οποία θα μπορούσατε να θεωρήσετε κατά κάποιο τρόπο ως κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στη συνέχεια ε, μελετώνται μέχρι την τελική έγκριση από τα δύο σώματα, από το Κοινοβούλιο, όπως είδαμε, το μόνο σώμα το οποίο εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες και αφετέρου το Συμβούλιο. Ονομάζεται και Συμβούλιο των Υπουργών, διότι εκεί συνεδριάζουν οι υπουργοί κάθε κράτους μέλους. Έτσι λοιπόν έχετε από τη μία πλευρά το Συμβούλιο, δηλαδή το σώμα που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις και αφετέρου από την άλλη πλευρά το Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Επαναλαμβάνω, αυτά τα δύο σώματα εργάζονται μαζί για την εκπόνηση νόμων, για την πρόθεση προτάσεων που βελτιώνουν όλο και περισσότερο την καθημερινή μας ζωή όπως γνωρίζετε καλά, είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν λειτουργεί πάντα τέλεια, πολλές φορές επικρίνεται, ωστόσο λειτουργεί. Είναι ένα μοντέλο που πολλές νέες δημοκρατίες ε, στις χώρες του τρίτου κόσμου προσπαθούν να μιμηθούν, διότι πρόκειται για την ύψιστη, δυνατή μορφή δημοκρατίας. Και πάντα στο όνομα αυτής της δημοκρατίας, στο Κοινοβούλιο, Αποφασίζει επίσης να προωθεί μια μεγάλη σειρά πρωτοβουλειών όπως αυτήν εδώ σήμερα, για την οποία συνεδριάζουμε σήμερα. Σήμερα, επαναλαμβάνω, έχετε ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών αρκετά εντατικό και αρκετά πυκνό. Γι' αυτό το λόγο δεν θα σας ε, απασχολήσω περισσότερο. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο, τον κύριο Κλάρκ, ώστε να κηρύξει επίσημα την έναρξη των εργασιών σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και σας εύχομαι μια εξαιρετική και επικοδομητική ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μάρκο. Πρέπει βέβαια να είμαστε νοικοκυρεμένοι εδώ. Πρέπει να φοράτε τα ακουστικά σας για να μπορείτε να παρακολουθείτε τη μετάφραση η οποία προσφέρεται σε όλες τις κοινοτικές ε, γλώσσες. Θα δείτε τους αριθμούς με τις γλώσσες στις καμπίνες μπροστά, οπότε ανάλογα προσαρμόζετε και το κουμπί των ακουστικών σας. Επίσης, ε, μπορεί να σας βοηθήσουν και πίσω στην αίθουσα, υπάρχουν ε, κλητήρες, ό,τι χρειάζεστε. Σήμερα θα δουλέψουμε μέχρι τις 12.30. Θα διακόψουμε στη συνέχεια για το γεύμα και θα συνεχίσουμε μετά από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ε, θα χωριστεί το πρόγραμμα σε, τρεις, ε, σε τρία κομμάτια. Πρώτα θα ασχοληθούμε με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και την εφαρμογή της στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Θα εξετάσουμε την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την εφαρμογή λοιπόν της σύμβασης αυτής στα πλαίσια της κρίσης. Θα συζητήσουμε στρατηγικές προκειμένου να βγούμε από την κρίση και τέλος στο τρίτο μέρος θα συζητήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων ε, με αναπηρίες, πώς θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια και θα επικεντρωθούμε λοιπόν στα δικαιώματα των πολιτών και την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια της ε, ε, πράξης για την προσβασιμότητα. Υπάρχει ένας κατάλογος ομιλητών προκαθορισμένος εδώ θα ακολουθήσουμε, όπως είπαμε, τους κανόνες που ισχύουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν συνεδριάζει σε Ολομέλεια. Θέλω όμω να υπογραμμίσω εδώ ότι όσοι έχουν χρόνο μιλία μπορεί να μην τον πάρουν ακριβώς τη στιγμή που το ζήτησαν. Το γεύμα θα λάβει η χώρα στο χώρο Μενουίν, που είναι ένας ανοιχτό χώρος που βρίσκεται στο ίδιο αυτοκτήριο, αλλά δύο ρόφους πιο κάτω προσφέρεται για όλους τους συμμετέχοντες και τους ευρωβουλευτές και όλους όσους βρίσκονται στην αίθουσα, εκπροσώπους των ευρωβουλευτών κλπ. Ο καφές, αν οπωσδήποτε θέλετε καφέ, σε μισή ώρα περίπου, τέλο πάντων στις 10 και 4 θα σερβιριστεί ο καφές. Στο τέλος, δηλαδή γύρω στις 5.30 θα ψηφίσουμε το ψήφισμα με μία ψηφοφορία, έτσι που ονομάζεται «Όραμα για την επόμενη δεκαετία», εφαρμόζοντας την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε καιρούς κρίσης. Το ψήφισμα αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας ε, των μελών εδώ. Πολλοί έχουν υποβάλει και τροπολογίες, έχουν κάνει σχόλια επί του ψηφίσματος αυτού που ελήφθησαν υπόψη στο κείμενο που έχουμε μπροστά μας. Η ψηφοφορία λοιπόν θα γίνει ε, πάνω στο ψήφισμα λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Φόρου Ατόμων με Αναπηρία. Να ξέρετε ότι αν θέλετε να βγάλετε φωτογραφίες χωρίς φλάς παρακαλώ και τα κινητά να ξέρετε ότι αν είναι ανοιχτά κάνουν παρεμβολές και υπάρχει πρόβλημα και με την ε, διερμηνία τότε. Οπότε σας παρακαλώ κλείστε τα κινητά σας. Πάντως όταν φύγετε από την αίθουσα ξανανοίξτε τα, μην το ξεχάσετε. Σύντομα τώρα θα σας παρουσιάσω το, την τελευταία εκδοχή του ψηφίσματος που τροποποιήθηκε όπως είπαμε βάσει των σχολείων που πήραμε από τους εκπροσώπους εδώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που βοηθήσατε να ενισχυθεί το κείμενο και να είναι πληρέστερο. Το ψήφισμα υπάρχει στα αγγλικά, στα γαλλικά και μπορείτε να το βρείτε και σε άλλη μορφή. Η τελική εκδοχή του ψηφίσματος θα αν ε, έχει μεταφραστεί από εσά και στις υπόλοιπες γλώσσες, παρακαλώ δώστε το στην ε, ε, γραμματεία για να μπορέσει να κυκλοφορήσει σε όλες τις γλώσσες. Υπάρχει και μεταγραφή του βέβαια. Θα γίνεται μεταγραφή όσο το διαβάζω. Καλύπτει διάφορες ε, πράξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αποτελείται από πέντε τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, τα μέτρα που πρέπει να λυθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να βγούμε από την κρίση, αναφέρεται η μεταρρύθμιση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες προκειμένου να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα κοινωνικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει στις αρχές της επόμενης χρονιάς ένα πακέτο για κοινωνικές επενδύσεις θα πρόκειται για παιδίσεις μακροχρόνιες και για μέτρα κοινωνική προστασίας που θα διασφαλίσουν την ζωή των ατόμων με αναπηρίες ως ανεξάρτητα άτομα. Θα επικεντρωνόμαστε στο θέμα των γυναικών, των νέων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες και την ε, φροντίδα τους. Λαμβάνεται υπόψη επίσης και η οικονομική πολιτική των χωρών ε, μελών και η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και λαμβάνονται υπόψη και συστάσεις για όλες τις χώρες προκειμένου να εντάσσονται καλύτερα στην κοινωνία τα άτομα με αναπηρία. Στο δεύτερο τμήμα ζητάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα ώστε να ε, φροντίσει για την ένταξη και όχι για τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρίες. Αναφέρονται διάφορα μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση υπέρ της προσβασιμότητας των ατόμων αυτών, υπέρ της καινοτομίας και των μεταφορών. Μιλάμε για τα διευθυντικά ταμεία εδώ, για την διευκόλυνση Connecting Europe που βοηθάει στις μεταφορές και μιλάμε και για ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα και για διεθνή συνεργασία. Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα που διαπραγματεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις μέρες. Στο τρίτο τμήμα μιλούμε για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εφαρμόσει την σύμβαση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων υπάρχει διαδικασία να διασφαλίσουμε ότι όλη η νομοθεσία συμμορφώνεται και δεν προβλέπει διακρίσεις, ε, τις συλλογικές συμβάσεις την πρόσβαση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των διαδικασιών πρόληψης υπέρ των ατόμων με αναπηρίες, δηλαδή να μην γίνεται διάκριση σε βάρος τους. Το τέταρτο σημείο μιλάει για την προσβασιμότητά μας. Η νομοθεσία για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, και για την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας. Είναι πράγματα τα οποία θέλουμε να δούμε στην τελική νομοθεσία. Υπάρχει επίσης ένα θέμα για μέτρα υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρίες, όπως επίσης και για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Τέλος, συμπεριλαμβάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις που θα ακολουθήσουν μετά τη συζήτηση αυτή. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζεται λοιπόν σε όλα αυτά και είναι η συνεισφορά μας στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της σύμβαση του ΟΗΕ. Η Ολομέλεια στην Ολομέλεια συμμετέχουν οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες. Task Force, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης για την εφαρμογή της ε, σύμβασης αυτή, που, της οποίας ηγείται η Επιτροπή Αναφορών. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άτομα με αναπηρίες ε, συμμετέχουν και σε κάθε εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προτείνουμε λοιπόν το ψήφισμα αυτό να εγκριθεί από το Σώμα στο τέλος. Τώρα το λόγο έχει ο Γιάννης Βερδικαστάνης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρου Ατόμων με Αναπηρίες. Γιάννη, έχεις το λόγο για να προεδρεύσεις ε, την ε, κήρυξη της έναρξης των εργασιών μας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο τρίτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία. Νομίζω ότι πριν ε, προχωρήσουμε στο official opening πρέπει να έρθει μαζί μας ο αξιότιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος ε, Σούλτς, ο οποίος αναμένεται νομίζω θα γυρίσω στα αγγλικά τώρα. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι τις 10 παρατέταρτο, μέχρι ότου αφηχθεί ο Πρόεδρος, για να γίνει και η επίσημη έναρξη. Θα πρέπει να, να ξεκινήσουμε... Πρέπει να πούμε ότι ξεκινήσαμε αρκετά γρήγορα, προχωρήσαμε και είμαστε πιο μπροστά από το χρόνο που είχαμε προβλέψει. Ας μείνουμε στην αίθουσα λοιπόν, περιμένοντας την άφηξη του Προέδρου για να γίνει η επίσημη έναρξη αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης σήμερα. Please, please. Πού είναι το. Ναι, κλειστά. Πού είναι το κουδούνι. Δεν κουδούνι. Χτύπησε το όπως το έκανε με το ανάποδο κάτω. Can you, can you hear me? Με ακούτε παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να, βάλε, να έχετε πάντοτε τα ακουστικά. Μόνο έτσι δουλεύει το σύστημα για να με ακούτε, να με καταλαβαίνετε. Σας παρακαλώ να μείνετε καθισμένοι στις θέσεις σας. Ανα πάσα στιγμή αναμένεται η άφηξη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ξεκινήσουμε αμέσω. Σας παρακαλώ να μείνετε στις θέσεις σας. Με πολύ υπομονή βέβαια. δεν έχει κανένα δεν έχει κανένα δεν έχει με δεν έχει you.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 Please take your seats. Please. Καθίστε παρακαλώ. And now... Τώρα Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε με την κήρυξη της έναρξης του Τρίτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άτομα με, των ατόμων μάλλον με αναπηρίες. Και είναι τιμή μας που έχουμε εδώ μαζί μας τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μάρτιν Σούλτς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πρώτη μέρα της ε, δημιουργίας του απετέλεσε έναν ισχυρό σύμμαχο και έναν ε, αξιόπιστο σύμμαχο και κάποιο όργανο που υποστήριξε πάρα πολύ τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι έπαιξε έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο νομοθετώντας υπέρ των ατόμων με αναπηρίες, με προγράμματα και με ψηφίσματα που θέλουν την ένταξη, τη μεγαλύτερη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία μας. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα περίπου 500 εκπρόσωποι ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες και των οικογένειών τους βρίσκονται εδώ επί τη ευκαιρία αυτή. Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή για μας που σας έχουμε μαζί μας για να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών μας. Έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο δικό σας οίκο, στο δικό μας, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. με κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί προσκεκλημένοι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που αισθάνομαι που μπορώ σήμερα να, να κηρύξω την έναρξη των εργασιών του Τρίτου Κοινοβουλίου για άτομα, των ατόμων με αναπηρίες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Βαρδακαστάνης με υποδέχθηκε με τα ευγενή του λόγια και τον ευχαριστώ θερμά ως Προέδρο του European Disabilities Forum και την κυρία Τζόρτζη την ε, Διευθύντρια του Φόρουμ αλλά κυρίως θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τους, ε, για τις ε, επίπονες προσπάθειες για την οργάνωση της παρούς εκδηλώσεως και σας ευχαριστώ θερμά για το πολύ επικοδομητικό πνεύμα που επιδείξατε κυρία Βαλτέζη σε αυτή την προσπάθεια. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία, το πνεύμα συνεργασίας που μας επέτρεψε να φτάσουμε στη σημερινή τρίτη αυτή εκδήλωση του Κοινοβουλίου των ανθρώπων με, των ατόμων με αναπηρίες. Πρόκειται για ακόμη ένα αποτέλεσμα της ε, δουλειάς μιας από τις παλαιότερες διακοινοβουλευτικές ομάδες που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή της ε, διακοινοβουλευτικής ομάδας για τα άτομα με αναπηρίες, μια ε, επαφή, ένας χώρος επαφής και επικοινωνίας των ευρωβουλευτών μας με την κοινωνία των πολιτών και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους δικούς μου βουλευτές, ε, συναδέλφους βουλευτές που συμμετέχουν στη διακοινοβουλευτική αυτή ομάδα και που βρίσκονται εδώ σήμερα βέβαια παρόντες. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας συνάντηση λαμβάνει η χώρα σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη διέρχεται το, τρίτο το πέμπτο έτος της. Η ανεργία έχει ανέβει κατά 11%. Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη είναι διπλάσια. Υπάρχουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν περιπέσει σε βαθύτατη ύφεση και η απάντηση που δίνουν πολλές εθνικές κυβερνήσεις στα προβλήματα αυτά είναι περικοπές άνευ προηγουμένου. Βεβαίω και χρειάζεται η δημοσιονομική πειθαρχία, η εξυγίανση δημοσιονομική καλύτερα. Εμεί, εγώ προσωπικώ, αλλά ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε σύμφωνοι με το στόχο των ε, ισοσκελισμένων προπολογισμών. Αλλά δεν μπορούμε να λησμονούμε, γιατί δεν μπορούμε να λησμονούμε τι επόμενε γενναίε, δεν μπορούμε δηλαδή να επιβαρύνουμε τι προσεχεί γενναίε με την ε, ευημερία τη δική μας με, τα, με τις δαπάνες της δικής μας για την διαβίωσή μας. Πλην όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί ότι η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι μονομερής, διότι καθίσταται σαφές και ξεκάθαρο πλέον ότι χωρίς ανάπτυξη δεν πρόκειται ποτέ να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία. Ταυτόχρονα πολλές περικοπές λαμβάνουν χώρα, περικοπές οι οποίες πλήττουν τους πιο αδύναμους στις κοινωνίες μας. Και έτσι προκύπτει σαφής κίνδυνος να οπισθοδρομήσει και η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και να φτάσει στην κατάσταση που είχαμε πριν από δεκαετίες ολόκληρες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κατά μέσον όρο πιο φτωχό το άτομο με αναπηρία από ότι ο μέσος πολίτης. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό εκείνων ε, που ζουν ε, κάτω από το όριο της φτώχειας, 21% λένε οι στατιστικές, ένα στους πέντε δηλαδή, ή ε, συνθήκες διαβίωσης, απασχόλησης σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό σε πολλά κράτη είναι χειρότερες. Αυτό βέβαια συνεπάγεται επιπλέον κόστος, όχι μόνο για τον ε, ίδιο τον άνθρωπο, για το ίδιο το άτομο με αναπηρίες, αλλά γενικότερα για την κοινωνία και πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται να βοηθείτε το άτομο με αναπηρίες και στην ε, αναζήτηση εργασίας Και πρέπει να πω ότι αυτό, εάν ε, θέλουμε να το δούμε και οικονομικά, είναι πολύ πιο συμφέρον για την, κοινωνία οικονομικά από ότι το να αποκλειστεί το άτομο αυτό και να μπει στο περιθώριο. Έχουμε λοιπόν δυσκολία ως προς την πρόσβαση και στο χώρο εργασίας αλλά και στην εκπαίδευση και είναι σαφές για μένα ότι η κοινωνία μας εν μέσω κρίσεως δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς τις δυνατότητες που έχουν τα άτομα με αναπηρία, το δυναμικό που προσφέρουν. Τι άλλο λοιπόν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να έχουμε γιατί υπάρχει ήδη τομεακή, τομεακού χαρακτήρα ε, νομοθεσία, παραδείγματι για τις αερομεταφορές που εγκρίνεται σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά ε, έχει ζητήσει και εγκρίνει μέτρα για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες ε, και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Πρόσφατα ακόμη με την οδηγία για την βελτίωση των δικαιωμάτων των θυμάτων ε, ποινικών αδικημάτων αποδείξαμε ότι είμαστε στο, στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την προστασία εκείνων που έχουν περισσότερο ανάγκη υποστήριξη. Επίσης, την υλοποίηση των ε, μέτρων που απαιτείται να λάβουν τα κράτη-μέλη Είμαστε, πρέπει να πω, το πρώτο, κοινοβούλιο που, έχει τον, που υποδέχθηκε το 2009 το Άνταμ Κόζα, τον κοφάλαλο συνάδελφο που όλοι γνωρίζετε ασφαλώς. Επίσης, στο κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως για το προσωπικό μας έχουμε συμπεριλάβει αντίστοιχες διατάξεις και τη δυνατότητα απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ε, παιδιών αυτών, αλλά και δυνατότητες ακόμη εξάσκησης με ε, ειδικέ συμβάσεις για άτομα με ειδικέ ανάγκες. Όλα αυτά όμως, ξέρετε, είναι μόνο κομμάτια ενός μοσαϊκού, ενός ευρύτερου μοσαϊκού που όμως δεν υπάρχει σαν γενικό όραμα. Γιατί πρέπει οι ανάγκες των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, οι απαιτήσει τους να ε, παρισφρήσουν σε κάθε τομέα δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα θέματα των μεταφορών μέχρι την πολιτική της συνοχής, από την έρευνα μέχρι την δημοσιονομική ε, πολιτική, μέχρι τον οικονομικό συντονισμό, μέχρι τις δημόσιες προμήθειες αλλά και την αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα των ατομών με αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα, όπως ίσως τα γνωρίζετε, αλλά και τα περισσότερα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής, της, ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέλη. Άπαξ λοιπόν και αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η σύμβαση και συμμετάσχει στην ε, υλοποίηση της και η κοινωνία των πολιτών θα μπορέσουμε πιστεύω να έχουμε μια ε, πραγματική διάσταση, ένα πραγματικό όραμα, αυτό το όραμα στο οποίο αναφέρθηκαν νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερως έχει προχωρήσει στην υποβολή μιας προτάσεως νομοθετήματος για τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ε, τη λεγόμενη δηλαδή European Accessibility Act, πράξη προσβασιμότητας. Πρόκειται για ένα μέσο νομοθετικό το οποίο καλωσορίζουμε φυσικά. Πιστεύουμε ωστόσο και προειδοποιούμε ότι θα πρέπει σε κάθε λεπτομέρεια αυτού του νομοθετήματος να γίνουν οι σωστές προτάσεις και μόνο όταν δούμε ότι είναι όλες οι προτάσεις σωστές σε κάθε σημείο του θα το εγκρίνουμε διότι νομοθετήματα τα οποία δεν είναι επαρκώς λεπτομερή για το ζήτημα αυτό για μας είναι ανεπαρκή και ατελή. Κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνοντας την παρούσα εκδήλωση νομίζω διακηρύσει την σαφή του υποστήριξη, εμπλοκή και συμμετοχή στα προβλήματα των ΑΜΕΑ. Είμαι προσωπικός πεπισμένος ότι ο βαθμός ανάπτυξης, εξέλιξης μιας κοινωνίας προσμετράται και πρέπει να προσμετράται από τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αυτή αντιμετωπίζει και προστατεύει τα πιο ευάλωτα μέλη της. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και για τη συνειδητοποίηση μέσα στην, ε, στις κοινωνίες μας και για την πρόσβαση στο χώρο εργασίας, στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στην, ε, κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, στην, στις υπηρεσίες υγείας. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν, τα όποια προσκόμματα υπάρχουν πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να αγωνιστούμε για την ε, κοινωνική ενσωμάτωση, για την αλληλεγγύη, διότι δυστυχώς αυτές οι έννοιες και αξίες δεν είναι αυτονόητες στις κοινωνίες μας. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλέ και επικοδομητικέ εργασίε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσε οι συζητήσει σα και ταυτόχρονα σα ζητώ συγγνώμη εάν δεν μπορέσω, γιατί δεν θα μπορέσω να παραμείνω και να συμμετάσχω σε όλη τη διάρκεια των εργασιών σας και είμαι εδώ παρόν μόνο για την κήρυξη της ενάρξεως, διότι σήμερα έχω να ε, επισκεφτώ και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι ο Πρόεδρος έχει το προνόμιο αλλά και το καθήκον να παρίσταται και να συντονίζει πολλές εκδηλώσεις ε, στο ε, κτίριό μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ, εάν βλέποντας ότι αποχωρώ μετά αυτά τα εναρκτήρια λόγια ε, εάν σας φανεί δυσάρεστο μην θεωρήσετε ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ασέβειας ή έλλειψη σεβασμού προς την εκδήλωσή σας. Είναι απλώς οι άλλες δεσμεύσεις μου που με υποχρεώνουν να αποχωρήσω. Σας ευχαριστώ. President. Κύριε Πρόεδρε, το γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι έχετε αναλάβει δέσμευση απέναντι στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Από τη δικιά μας την πλευρά, στο δικό μας τον αγώνα, ξέρουμε ότι έχουμε και εσάς μαζί μας για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα κρίσης. Όλα αυτά που είπατε ισχύουν. Εμείς αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι οι υποχρεώσεις που έχετε, οι ανηλυμένες, ε, σας αναγκάζουν να αποχωρήσετε. Γνωρίζουμε όμως ότι στο πνεύμα θα βρίσκεστε ακόμα μαζί μας ολόκληρη την ημέρα. Εκ μέρους όλων μας θέλω προσωπικά να σας ευχαριστήσω για την ε, δέσμευση που έχετε αναλάβει απέναντί μας, για την στήριξη που μας έχει προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές οι οποίοι έχουν στηρίξει την παρουσία όλων σχεδόν των εθνικών αντιπροσωπιών εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσία σας και προσβλέπουμε σε μια καρποφόρα συνεργασία μεταξύ μας μέσα σε αυτούς τους τόσο ταραγμένους καιρούς γεμάτους προκλήσεις για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Thank Ladies uh, Κυρίες και κύριοι, διακεκριμένοι, προσκεκλημένοι και συμμετέχοντες, ε, σας καλωσορίζω όλους στο τρίτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα άτομα με αναπηρίες. Ιστορική εκδήλωση σε ταραγμένους ε, Ιστορική σημασία καιρό. Το ευρωπαϊκό κίνημα για τα άτομα με αναπηρίες σήμερα σε αυτή την εντυπωσιακή συγκέντρωση θα συζητήσει και θα συμφωνήσει μια στρατηγική για τα επόμενα χρόνια. Τα δύο προηγούμενα κοινοβούλια για άτομα με αναπηρίες έλαβαν επίσης χώρα σε ζωτική σημασία, στις ιστορικές ε, στιγμές. Η πρώτη έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 1993 καθοδηγήθηκε από την DPI. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς εκείνους που μπόρεσαν να συμμετέχουν σε εκείνη την εκδέλωση. ιστορική σημασίας διότι έλαβε χώρα κατά την πρώτη ευρωπαϊκή ημέρα για τα άτομα με αναπηρία το Δεκέμβριο του 1993. Εκείνη τη χρονιά επίσης ε, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τους ε, κανόνες ίσων ευκαιριών για άτομα με αναπηρίες των Ηνωμένων Εθνών. Η δεύτερη έλαβε χώρα το 2003, το ευρωπαϊκό έτος για άτομα με αναπηρίες. Και τώρα η σημερινή εκδήλωση. Οι δύο προηγούμενες εκδηλώσεις δημιούργησαν μια ορμή όσον αφορά τα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Αναμφίβολα έχει σημειωθεί πρόοδος. Σε πολλούς τομείς Πασχόληση, κοινωνική προστασία, νέες τεχνολογίες σε διάφορους τρόπους μεταφορών, διαρθρωτικά ταμεία, κρατικές ενισχύσεις, δημόσιες συμβάσεις, ανθρώπινα δικαιώματα. Για να αναφέρω απλά μερικούς. Αλλά επίσης αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα σε αυτή την ταραγμένη εποχή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέτος είναι πιθανώς ε, η σημαντικότερη από τις τρεις εκδηλώσεις και περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. Σήμερα στην Ευρώπη διερχόμαστε ε, μέσα από τις χειρότερες ε, υφέσεις πότε όσον αφορά δικαιώματα για τα οποία πολεμήσαμε για πολλές δεκαετίες ποτέ στην ιστορία τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία δεν αναγνωρίζονταν καλύτερα σε νομικές διατάξεις και στις πολιτικές συζητήσεις και ποτέ στην πρόσφατη ιστορία δεν βρεθήκαμε υπό τόσο μεγάλη απειλή λόγω της ύφεση και της ε, δράσης, της απευθείας δράσης κατά των δικαιωμάτων μας λόγω μέτρων που έχουν ληφθεί από κράτη-μέλη με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν όχι σε κάθε περίπτωση τις περισσότερες οι πολιτικοί της Ευρώπης δεν έχουν κάποιο σαφές συνεκτικό σχέδιο, κάποια στρατηγική για να μας βγάλουν από αυτή την κρίση. Δεν υπάρχει κοινή συμφωνία για κατάλληλα μέτρα τα οποία θα χρειαστεί να ληφθούν ώστε να προστατευτούν τα άτομα με αναπηρίες από μια κρίση που όπως είπα νωρίτερα ε, είναι μια κρίση για την οποία δεν ευθύνονται. Το παρόν κοινοβούλιο είναι ένας τρόπος για να δείξουμε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μία μόνο μπορεί να είναι η απάντηση για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίσιμη σημασίας κατάσταση. Η απάντηση αυτή είναι απλή είναι σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη συμμετοχή και πιο ενοποιημένες δράσεις από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Εντολής και της προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα, εδώ, είμαστε περισσότεροι είμαστε ισχυρότεροι, θα χρειαστεί να ακουστούμε και πιο δυνατά. Βρισκόμαστε στον οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε τα δικαιώματά μας. Είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε να είμαστε παρόντες όταν λαμβάνονται αποφάσεις να διεκδικήσουμε να ακουστεί η φωνή μας. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω, πριν μιλήσω για το μέλλον, για να θυμηθούμε εκείνους μεταξύ μου, τους πιο ευάλωτους, κυρίως τις γυναίκες με αναπηρίες, τους νέους με αναπηρίες, παιδιά με αναπηρίες. άτομα με αναπηρίες που χρειάζονται υποστήριξη ψηλού επίπεδου. Και φυσικά θα πρέπει όχι μόνο να θυμόμαστε, αλλά να δράμε, ώστε να προστατεύουμε τους συναδέλφους μας, τους συναδέλφους μας εκείνους που εξακολουθούν να ζουν σε ιδρύματα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε με τη δική μας φωνή. χωρίς ενδιάμεσους. Χωρίς εξωτερική συμμετοχή. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τους ευρωβουλευτές. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα αποτελέσει φάρο για τις δράσεις μας στο μέλλον. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να προσφέρει τις κατευθύντηρες γραμμές για όλους τους ενδιαφερομένους στους τομείς των ατόμων με αναπηρίες για την επόμενη δεκαετία. Χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο για την Ευρώπη, για τους ανθρώπους με αναπηρία. Η κρίση έχει συνθλίψει όλες τις προσπάθειες που είχαν σχεδιαστεί, όλα τα προγράμματα, τα σχέδια, τις ιδέες, τις στρατηγικές που υιοθετήθηκαν στο παρελθόν, ακόμη και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Όλες αυτές οι στρατηγικές είναι ήδη απερχαιωμένες. Σήμερα η Ευρώπη είναι διαφορετική και στο μέλλον θα αλλάξει ακόμη περισσότερο, στο εγγύς μέλλον. Οι παλιές συνταγές λοιπόν δεν θα φέρνουν πλέον αποτελέσματα. Το σχέδιο για την Ευρώπη και τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές όλοι οι ευρωπαϊκοί νόμοι πρέπει να είναι συμβατοί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες. Κανένα ευρώ δεν πρέπει να δαπανάτε σε δομές, σε υποδομές χωρίς πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητα το European Accessibility Act, θα πρέπει να είναι μια πραγματική πράξη που θα παράσχει πραγματική προσβασιμότητα σε εικονικά, πραγματικά, φυσικά περιβάλλοντα, σε αγαθά και σε υπηρεσίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σλόγγαν «Τίποτα χωρίς, ε, για εμάς χωρίς εμάς», όπως συνηθίζω να ε, λέω, δεν είναι απλά ένα σλόγγαν, είναι ένας τρόπος ζωής για εμάς. Σε αυτές τις εποχές κρίσης, που στερούν δικαιώματα, υπηρεσίες, που στερούν την καρδιά του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, το ευρωπαϊκό κίνημα για άτομα με αναπηρίες, ενωμένο, δυνατότερο, θα συνεχίσει να αγωνίζεται, να προστατεύει και να προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. είναι ύψη τη σημασία, Αυτή η συνεδρίαση να μας οδηγήσει τα πίσω στις χώρες μας αποφασισμένους. Αποφασισμένους να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας από τα μέτρα λιτότητας που αποτελούν άμεσες παραβιάσεις και καταχρήσεις των δικαιωμάτων που έχουν προβλεφθεί στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες. Εγώ έχω την τιμή και μια ιστορική ευκαιρία την Κυριακή αυτή να βρεθώ στη Μαδρίτη σε μια εντυπωσιακή διαδήλωση που οργανώνεται από, την, από το Ισπανικό κίνημα για άτομα με αναπηρίες όπως κάναμε και στην Ελλάδα Γνωρίζω στην Πορτογαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία και σε πολλές άλλες χώρες. Χρειάζεται οι δράσεις μας να γίνουν πιο ριζοσπαστικές. Σας ευχαριστώ λοιπόν ξανά για την παρουσία σας. Σας εύχομαι σε όλους, σε όλους μας η εκδήλωση σημερινή να είναι επιτυχής. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βατρώνη. Τσόνη, πρόεδρο της ε, Επιτροπής ε, Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα προεδρεύσει την πρώτη ολομέλεια. Τίποτα για μας, χωρίς εμάς, χωρίς τη συμμετοχή μας. Πείτε το, μέχρι τα χωριά, μέχρι τις κομοπόλεις, μέχρι τις πόλεις, στις καρδιές όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία αλλά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε και εμείς να καλωσορίσουμε πλευράς μας την ε, ε, όλους εδώ τους παρισταμένους για την παρουσία τους εδώ και ξεκινάμε τις εργασίες μας για τα θέματα της νομοθεσίας και της υλοποίησης της ε, νομοθεσίας για τα άτομα με ε, αναπηρίες εν ώψη της οικονομικής κρίσης. Η κυρία Ματσόνη θα προεδρεύσει στο πρώτο αυτό τμήμα της συστήσεως, αλλά πρώτα θα πρέπει νομίζω να πω εγώ δύο λόγια για, το, για την εκδήλωσή μας. Θα μιλήσουμε για την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως είπα, κατά τη διάρκεια αυτής της ολομέλειας. Εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε νομοθεσία που υιοθετήθηκε το, το 2006 με τη σύμβαση στην οποία κατέληξε η ε, Γενική Συνέλευση των Εθνών, μία σύμβαση η οποία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οδήγησε στην σύμβαση με 106 συμβαλόμενα μέρη που έχει σε συνέπεια να εφαρμόζεται ένα κείμενο σύμβασης στο οποίο έχουν συμπράξει και τα οι ίδιοι εμπλεκόμενοι, δηλαδή τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε είτε με σωματική αναπηρία, είτε με πνευματικά, ε, πνευματικές ελλείψεις ή καθυστερήσεις, με τα εμπόδια ως προς την ε, συμμετοχή στην κοινωνία που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες. Θεωρείται λοιπόν ε, σημαντική αξία η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στις κοινωνίες και ξέρουμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην ε, πολιτική διαδικασία από το στάδιο της σχεδίασης μέχρι την απτή διατύπωση της νομοθεσίας και την παρακολούθηση της υλοποίησής της στη συνέχεια. Πρέπει δηλαδή τα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν σε ολόκληρη τη διαδικασία και πρόκειται για μια συνθήκη, για μια σύμβαση την οποία για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε ως σύνολο. Όπως και κάθε επιμέρους κράτος μέλος τα 24 για την ακρίβεια, ενώ έχουν υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη, έχουν κυρώσει τα 24 από αυτά και έχει δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υλοποίηση αυτή τη σύμβαση και στην εξασφάλιση του ότι τα άτομα με αναπηρίε ε, θα έχουν ε, και οι προοπτικέ του θα ενσωματώνονται σε κάθε τομέα πολιτική. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσαρμόζεται δηλαδή κάθε τομέα της πολιτικής όπου έχει αρμοδιότητες και εξουσίες η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επιταγές αυτής της σύμβασης και επαληθεύεται η σχετική προσαρμογή. Χρειάζεται βέβαια πολλή δουλειά ακόμη. τόσο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, αλλά και άλλα πολιτικά σώματα, Φερρυπίν, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών κτλ. Ακόμη πολλή δουλειά μέρη να γίνει, διότι είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουν όλοι μαζί και να εξασφαλίσουν ότι θα επιφέρει πραγματική αλλαγή, πραγματική βελτίωση στις ζωές των ΑΜΕΑ η νομοθεσία. Η υλοποίηση αυτής της σύμβασης ε, προχώρησε την ε, τον προηγούμενο μήνα με την δημιουργία της Επιτροπής Εποπτείας ή Παρακολούθησης και έτσι θα έχουμε συνεργασία με την Επιτροπή των Αναφορών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και την Υπηρεσία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην εποπτεία αυτής της, ε, της εφαρμογής αυτής της συμβάσεως, ώστε να προσφέρεται και το κατάλληλο δυναμικό, αλλά και οι κατάλληλοι πόροι οικονομικοί και άλλοι στην Επιτροπή αυτή για να επιτελέσει το έργο της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει έκθεση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναφυπηρίες, όπως έχει προγραμματιστεί. Μια έκθεση πολύ σημαντική, μια έκθεση η οποία πιστεύουμε θα ε, ρίξει φως στο ζήτημα της καταγραφής της καταστάσεως αλλά και της καταγραφής των προόδων που έχουν επιτευχθεί εντωμεταξύ. Και έτσι μπορεί να αποτελέσει τον πρώτο θεμέλιο λίθο ενός προγράμματος δράσεως για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν σε επίπεδο κρατών μελών, είναι δυνατό να αξιοποιηθεί ως επιχείρημα η οικονομική κρίση για να ε, αποφύγει κανείς την υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση. Έχουμε αγωνιστεί όλοι πολύ σκληρά για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα της σύμβασης, αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Και γι' αυτό μιλούμε για ουσιαστική βελτίωση και στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και για δικαιώματα που έχουν τα ΑΜΕΑ για ιδιαίτερη υποστήριξη και βοήθεια και είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε για να διαφυλάξουμε αυτά τα δικαιώματα. Υπό το φως της συμβάσεως σκοπεύουμε να τα αναπτύξουμε περαιτέρω. Ιδιαίτερα πρέπει να ε, δώσουμε προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν αμαία ε, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης γιατί πρέπει να εξετάζεται τι είδους επιπτώσεις έχει η οικονομική κρίση στα νέα, στην απασχόλησή τους, στα, ε, στην εκπαίδευσή τους, στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες. Και αυτό με στόχο βέβαια να εξασφαλίσουμε την πλήρη ε, συμμετοχή τους στις κοινωνίες, την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων τους. Βλέπουμε ότι δυστυχώς υποφέρουν πρώτα από την οικονομική κρίση και άρα για να υλοποιηθούν οι στόχοι της Συμβάσεως των ΕΕ πρέπει να προσφέρουμε λύσεις για την καταπολέμηση του αποκλεισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό έχει πρωτο, πρωταρχικό ρόλο να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχάς ο συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση, αλλά και γιατί όπως σε ολόκληρο τον κόσμο έτσι και ειδικότερα στην Ευρώπη όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούνε πώς χειρίζεται τα θέματα αυτά, πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ. Με αυτά τα λόγια λοιπόν θα παρακαλέσω τη Ρομπέρτα Αντζελίν λάβει το λόγο, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ευχαριστώ που βρίσκεται μαζί μας και την παρακαλώ να λάβει το λόγο σύντομα για μία παρουσία στο αυτό. Ε, Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε που διοργανώσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη συνάντηση, την τόσο σημαντική συνάντηση με τόσου πολλού συμμετέχοντε. Ήθελα να σα καλωσορίσω ω αντιπρόεδρο. Ε, επιφορτισμένη με τα δικαιώματα των ε, νέων ε, σε αυτή την ομάδα εργασίας ασχολούμαστε με τις ίσες ευκαιρίες και με τις ε, επωνομαζόμενες διαφορές. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα Σημαντικό είναι να, που λαμβάνει η χώρα μια τέτοια εκδήλωση εντός των θεσμικών οργάνων ώστε να γιορτάσουμε τη Διεθνή ημέρα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το να τη γιορτάζουμε σε έναν τέτοιο χώρο σημαίνει ότι διατηρείται η επικέντρωση σε αυτά τα θέματα, στα προβλήματα αυτά, στις πιθανές ευκαιρίες. Έτσι, ευαισθητοποιούμε όλα τα θεσμικά όργανα, τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά θεσμικά όργανα και την κοινή γνώμη όσον αφορά τις στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν, οι βέλτιστες πρακτικές, αλλά και για να υπογραμμίσουμε τη σπουδαιότητα των αξιών, της αξιοπρέπειας, της ευημερίας των ατόμων με αναπηρίες, των ε, ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζήτημα που αφορά υπηρεσίες, προϋπολογισμό, συγκεκριμένα εργαλεία. Είναι και ζήτημα αξιών, διότι η διαφορετικότητα είναι μια αξία. Εγώ πιστεύω ότι τα άτομα με αναπηρίες ε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως άτομα με διαφορετικές ικανότητες. Δηλαδή εξίσου ικανα, ικανά άτομα με όλους τους υπόλοιπους με διαφορετικές απλά ικανότητες. Προφανώς τα άτομα αυτά με τις διαφορετικές ικανότητες θα πρέπει να απολαμβάνουν συνθήκες τέτοιες που να τους επιτρέπουν ίση, ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, στην εργασία. Πρέπει να τους δίνουμε την ευκαιρία να απολαμβάνουν ίδιες ευκαιρίες, ίσες ευκαιρίες. Διότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Εξάλλου, τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη ανέρχονται σχεδόν στο 80 εκατομμύρια πολύ σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων πολιτών. Δεν αποτελούν εξαίρεση. Δεν είναι μια μικρή μειονότητα. Είναι πάρα πάρα πολλοί πολίτες. Πρέπει λοιπόν να υπερασπιστούμε την έννοια, την αξία των ίσων ευκαιριών και την έννοια και την αξία της προσβασιμότητας. Προσβασιμότητα δεν σημαίνει μόνο να καταργούμε τα αρχιτεκτονικά προσκόμματα αλλά και όλα τα υπόλοιπα την έλλειψη υπηρεσιών την έλλειψη πολιτικών επαρκών μέτρων καθώς και των προκαταλήψεων. Ακόμη και οι προκαταλήψεις αποτελούν προσκόμματα για τα άτομα με διαφορετικές ικανότητες. Όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ότι μόνο το 5% των δημόσιων ιστοτόπων στα 27 κράτη-μέλη συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα προσβασιμότητας. Οι δημόσιες λοιπόν υπηρεσίες που είναι υπηρεσίες για όλους, για κάποιον, με διαφορετικές ικανότητες, είναι προσπελάσιμες μόνο εν μέρη μόνο το 5% αυτών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαρίθμησε ορισμένα από τα μέτρα τα οποία εμείς υιοθετούμε αυτή τη στιγμή εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε οι εργαζόμενοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με διαφορετικές ικανότητες να απολαμβάνουν αυτές τις προσαρμογές ώστε να μπορούν να εργάζονται ελεύθερα και με πλήρη προσβασιμότητα. Προσπαθήσαμε να εξαλείψουμε όλα τα εμπόδια του ίδιου του κτηρίου, οι ανελκυστήρες, τα γραφεία στην είσοδο να προσφέρουν δυνατότητες πρόσβασης ακριβώς τα άτομα με αναπηρία. Το κυριότερο όμως είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δεσμευτεί ώστε να καταφέρει συντονισμό και των 27 κρατών μελών για την εφαρμογή πολιτικών στο ύψος των προκλήσεων, των εξαιρετικά δύσκολων προκλήσεων που δυστυχώς επιδεινώνονται από την οικονομική κρίση. Καταλήγοντας στο συμπεράσματά μου, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα από τα προβλήματα που με απασχολεί περισσότερο το πρόβλημα των παιδιών με διαφορετικές ικανότητες. Στην Ευρώπη υπάρχουν σχεδόν 15 εκατομμύρια παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι πάρα πολλά 15 εκατομμύρια παιδιά. Παιδιά μεταξύ 16 και 19 ετών όπου το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου ισούται με 40%. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για παιδιά που πραγματικά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδείας, που συνεπώς εγκαταλείπουν το σχολείο, εγκαταλείπουν το, την παιδεία και καταλήγουν ενήλικες καταδικασμένοι στην ανεργία και στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε στη διαθεσή μας μαθαίνουμε ότι το ποσοστό ένδυας μεταξύ ατόμων με αναπηρία είναι άνω του 70% σε σχέση με το μέσο όρο των υπολείπων πολιτών. Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι αποκλεισμός των παιδιών από την πρόσβαση στο σχολεία, στην παιδεία, σημαίνει καταδίκη τους σε ένδια. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα σε αυτές τις περίοδους κρίσης. Το αποδεικνύει και μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Η γενική αίσθηση είναι ότι οι διακρίσεις στις αγορές εργασίας για λόγους αναπηρίας σημειώνει ισχυρή αύξηση κυρίως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν που διοργανώσατε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αληθινά τα άτομα με διαφορετικές ικανότητες δεν μπορούν να πληρώνουν αυτές το υψηλότερο τμήμα, τίμημα της οικονομικής κρίσης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να δεσμευτούν ώστε να διαφυλάξουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να μην αφήνουν πίσω, να μην παραμελούν, να μην εγκαταλείπουν κυρίως όσους χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντζελίνη, για τόσα μας είπατε. Και πιστεύω ότι από αυτά που είπατε μπορώ να πω ότι συμφωνείτε απόλυτα μαζί μας για το ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παιδεία, η εκπαίδευση και ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτήν. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό για να βρουν δουλειά στο μέλλον τα άτομα με αναπηρίες και να μην καταλήξουν στην ένδια. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα θέλω να δώσω το λόγο στην Συμπρόεδρο, την Εμίλια Ματσόνη. Η Εμίλια Ματσόνη είναι η Πρόεδρος της ε, Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδια για τις αναφορές. Πολύ σημαντική για μας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ σε αυτήν την τόσο σημαντική συνάντηση. Πρέπει να σας πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που έχω την ευκαιρία να πάρω το λόγο σε ένα τέτοιο σώμα και για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως είναι το θέμα των ατόμων με αναπηρίες που, είναι, που έχει κεντρική σημασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για μένα προσωπικά επίσης αλλά και ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών όπως είμαι. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιμονή σας. Στην αρχή είχαμε κάποιες δυσκολίες με την οργάνωση της συνάντησης αυτής και μόνο χάρη στη δικιά σας επιμονή καταφέραμε τελικά να την οργανώσουμε. Να οργανώσουμε δηλαδή αυτό το φόρουμ και έτσι να βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ σήμερα. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο βασικό βήμα έγινε με τη συνθήκη του Άμστερνταμ διότι εκεί στο άρθρο 13 η εισήχθη υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει τα άτομα με αναπηρίες από κάθε είδους διάκριση. Στη συνέχεια, υπογράφοντας και κυρώνοντας την σύμβαση του ΟΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε, μόνο πρόσθεσε κάποιες νέες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Και πρώτα απ' όλα την υποχρέωση να καταργήσει τα εμπόδια που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Στη συνέχεια είχαμε την δεκαετή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες που συμπλήρωσε το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τώρα με τη σύμβαση του ΟΗΕ, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Μεταφορών εντοπίζεται ως μέρος του ευρωπαϊκού πλαισίου όπως επίσης και ο Ευρωπαίος Συνήγορος του Πολίτη, ο Διαπεσολευητής... η Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αναπηρίες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, η Επιτροπή μας, η Κοινοβουλευτική Αναφορών, έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και είναι να προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η Κοινοβουλευτική αυτή Επιτροπή ε, συνεισφέρει και παρεμβαίνει κάθε φορά που χρειάζεται προστασία των ατόμων με αναπηρίες, δηλαδή κάθε φορά που παραβιάζουν τα κράτη-μέλη την σύμβαση αυτή του ΟΗΕ. Εμείς δεχόμαστε αναφορές από τους πολίτες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοιου είδους παραβιάσεις και για αποφάσεις που γενικότερα μπορεί να τους πλήττουν. Αναφερόμαστε συνεχώς έχουμε σαν σημείο αναφοράς μας δηλαδή την σύμβαση αυτή του ΟΗΕ. Είτε έχουμε εκθέσεις, είτε εκθέσεις πρωτοβουλίες, είτε ετοιμάζουμε newsletters, είτε επικοινωνούμε με τον τύπο κτλ. Τα άτομα με αναπηρίες μας ενημερώνουν και σε καθημερινή βάση διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ένα σώρο εμπόδια τα οποία τους εμποδίζουν να χαρούν πλήρως των δικαιωμάτων τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν προβλήματα για πρόσβαση στην απασχόληση, στις δημόσιες μεταφορές κλπ. κλπ. Τέτοιες αναφορές λοιπόν μας κάνουν να στραφούμε στους αρμόδιους φορείς και να επιζητήσουμε λύση. Είμαστε λοιπόν δεσμευμένοι για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των, ατόπων, των ατόμων με αναπηρίες Επίσης καταπολεμούμε κάθε διάκριση που γίνεται και κάθε παραβίαση που γίνεται των ε, νόμων ή των συμφωνημένων. Το 2009 πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα υπέγραψαν μία αναφορά που πήραμε που κατήγγειλε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Έτσι και εμείς πιέσαμε το Συμβούλιο να υιοθετήσει την οδηγία κατά των διακρίσεων που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες να μην αντιμετωπίζουν διακρίσεις όταν πρόκειται για την κοινωνική προστασία και να μπορούν να έχουν ε, απρόσκοπτα πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση. Όσον αφορά τώρα την χρήση των κονδυλίων από τα διαφορετικά ταμεία, Πρόσφατα λάβαμε μία αναφορά η οποία ε, καταδεικνύει ότι γίνεται κακή χρήση των κονδυλίων από τα διευθυντικά ταμεία από ορισμένε χώρες μέλη που έχουν επενδύσει τέτοια κονδύλια με μη ορθό τρόπο. Τα διορθωτικά ταμεία εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται για να στηρίζουν την ε, ανάπτυξη υπηρεσιών και υπέρ της συνειδητοποίησης για να προσφέρει δηλαδή στα άτομα με αναπηρίες και να ενισχύσει στρατηγικές υπέρ τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ότι η πρόταση για έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για τα στρατιωτικά ταμεία για την περίοδο 2014 με 2020 περιλαμβάνει μια διάταξη που αναφέρεται στις αναπηρίες και λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε πρόγραμμα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει δηλαδή ένα mainstreaming, δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη το θέμα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα προγράμματά της. Μία άλλη αναφορά αναφέρεται στην περίπτωση Lucy's Case και έχει να κάνει Πρόκειται για έναν πολίτη ε, του Ηνωμένου Βασιλείου που πήγε σε μια άλλη χώρα και δεν μπορεί να πάρει επιδόματα και λοιπά το άτομο αυτό στην χώρα που έχει εγκατασταθεί. Δεν του το επιτρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι Βρετανικές αρχές που το εμπόδισαν επειδή πήγε και εγκαταστάθηκε στην Ισπανία με την οικογένειά του. Εδώ ζητήσαμε ε, προδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2009 το ζητήθηκε αυτό και το 2011 απάντησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ότι κάτι τέτοιο μόνο μπορεί να ισχύσει σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στο κοινωνικό σύστημα. Εμείς στηρίξαμε ότι από την αρχή έπρεπε να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος με το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελικά Ήρθε ο αναφέρον στην Επιτροπή μας και παρουσίασε το θέμα, το εξήγησε στην Επιτροπή μας και ήταν εκεί και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή μας επέμεινε ότι βάσει της απόφασης που μιλάει για τη δυνατότητα εξαγωγής τέτοιων επιδομάτων, μια τέτοια απόφαση πρέπει να ισχύσει και στην περίπτωση της κυρίας Λούση Στιούαρτ. Ένα άλλο θέμα που είχαμε στην Επιτροπή μας είχε να κάνει με την πρόσβαση σε βιβλία και άλλα έντυπα Πρόκειται για άτομα με δυσλεξία ή με άλλες αναπηρίες που βρέθηκαν στην Επιτροπή μας. Και εμείς ε, επιμείναμε ότι πρέπει να υπάρξει μια διεθνής σύμβαση ώστε να υπάρξει και εξαίρεση για το copyright σε άτομα που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες αναπήρων. Οι αναφέροντες ήρθαν στην Επιτροπή μας, ε, τους ακούσαμε, ε, δείξαμε ότι καταλαβαίνουμε πολύ καλά τα προβλήματά τους και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε για μια δεσμευτική σύμβαση. Επίσης ζητήσαμε και διευκρίνηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο και συνεχίσαμε διαδικασίες για μια δεσμευτική σύμβαση και με άλλες μεθόδους όπως είναι οι προφορικές ερωτήσεις κλπ. Πήραμε θαραλέα απάντηση από τον Επίτροπο Μπαρνιέ, ο οποίος είπε ότι δεσμεύεται πλήρως για μια νέα προσέγγιση προς μια δεσμευτική σύμβαση και είναι έτοιμος να μιλήσει με όλες τις χώρες μέλη ατομικά με την καθεμία. Έχουμε και δραστηριότητες για γνωμοδοτήσεις, για εκθέσεις και για εκθέσεις πρωτοβουλίας. Και θα σας αναφέρω εδώ τη γνωμοδότηση που είχαμε για μια έκθεση που αναφέρεται στα δικαιώματα ε, και για τα δικαιώματα των πολιτών μέχρι το 2020 που μιλάει για καλύτερη αναγνώριση της σύμβασης για άτομα με αναπηρίες έτσι ώστε να μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στις ηθίκες και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις. Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων μόλις αυτή τη βδομάδα. Όσον αφορά τώρα την κρίση. Συμφωνώ με αυτό που ακούσαμε πριν, ότι η κρίση και οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια αυτής της κρίσης κινδυνεύουν να αποδυναμώσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Σε πολλές περιπτώσεις στην πραγματικότητα τα μέτρα λιτότητας μας πάνε πίσω όσον αφορά τα κοινωνικά επιδόματα που καθυστερούν για παράδειγμα πάρα πολύ. Η κρίση δυστυχώς εμποδίζει τα κράτη-μέλη από το να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα υπέρ των ατόμων με αναπηρίες. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αναθεωρήσουν την κοινωνική τους πολιτική και να φροντίσουν για συστήματα κοινωνικής προστασίας και για προγράμματα μείωσης της ένδυας. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται διαρθρωτικές ε, αλλαγές στα διάφορα συστήματα συντάξεων, για παράδειγμα, επιδημάτων. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρίες να είναι αυτόνομα, να μπορούν να δουλέψουν, να ταξιδέψουν, να συνεισφέρουν δηλαδή στο κάτω-κάτω στην ε, κοινωνία και στην μείωση του κόστους. Τα κράτη-μέλη πρέπει να οργανώσουν ε, τις μεθόδους τους με εξαιρέσεις, να φροντίσουν για την διαβίου κατάρτιση για τα άτομα με αναπηρίες στα πλαίσια του δυνατού. Τα κράτη-μέλη πρέπει επίσης να ενημερώνουν τα άτομα με αναπηρίες για τα θέματα που τους αναφέρουν. Η γενική αντίληψη όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες επίσης πρέπει να αλλάξει, νοτροπία δηλαδή. Και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε σε δράσεις και στρατηγικές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση για έναν κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνω. Λοιπόν, η πρόταση για έναν κανονισμό όσον αφορά τα διαφορετικά ταμεία για την περίοδο 2014 με 2020 περιλαμβάνει, λέω, μια διάταξη που βάζει εξάντε προϋποθέσεις για κάθε πρόγραμμα προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τα άτομα με αναπηρίες. Εμείς το υπογραμμίζουμε αυτό το σημείο. Γιατί πιστεύω ότι αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία και συνάδει με τους στόχους μας. Εν κατακλείδη, πιστεύω ότι πετύχαμε πολλά για τα άτομα με αναπηρίες κατά τον προηγούμενο αιώνα, όπως είπατε, αλλά νομίζω ότι παραμένουν ακόμα περισσότερα να γίνουν. Συμφωνώ λοιπόν με το ψήφισμά σας και θα στηρίξω τα πέντε αιτήματά σας, που αναφέρονται δηλαδή στο ψήφισμα. Ιδιαίτερα πιστεύω ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία στα πλαίσια ακριβώς του ΟΗΕ και της σύμβασης αυτής, έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα νέο κοινωνικό μοντέλο για τα κράτη-μέλη, για να εφαρμοστούν θέματα που έχουν να κάνουν με θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα την ελευθερία μετακίνησης και προκειμένου να πιέσουμε ώστε να εγκριθεί η οδηγία κατά των διακρίσεων. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ. Κύριε Ματσόνη, ασφαλώς και θέλουμε και στηριζόμαστε στη συνεργασία μαζί σας και για το μέλλον, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρακολούθηση των... της νομοθεσίας. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο, τον διαμεσολαβητή, Ευρωπαίο διαμεσολαβητή, εκφράζοντας τη χαρά μου για την αποδοχή από πλευρά της προσκλήσεως για συμμετοχή στην συνέλευσή μας, στη συνάντησή μας. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει ο ίδιος εδώ, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα για μία βίντεο διάσκεψη. Θα τον δούμε από μακριά, τον κύριο Διαμαντούρο, και θα συνομιλήσουμε μαζί του. Σας καλωσορίζω, κύριε Διαμαντούρο. Σας ευχαριστώ, κύριε Διαμαντούρο. Και θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε εκφράζοντας τη χαρά μας που έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στην εκδήλωσή μας, έστω και αν σας βλέπουμε μόνο από βίντεο διάσκεψη. Σας δίνω λοιπόν το λόγο αμέσως. Υποθέτω ότι μου έχετε δώσει το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Σωστά. Ωραία, ευχαριστώ. Αξιότιμη Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, αξιότιμη Πρόεδρε του Φόρουμ του Ευρωπαϊκού για τα άτομα ε, με αναπηρίες, κύριε Βαρτακαστάνη αξιότιμα μέλη του φόρου, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να αρχίσω εκφράζοντάς σας τις θερμές μου ευχαριστίες. Καταρχήν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρίες που με προσκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που με προσκαλέσατε λοιπόν να έρθω και να είμαι μαζί σας επί τη ευκαιρία αυτή. Φυσικά θα είχα προτιμήσει να βρίσκομαι όντως ε, μεταξύ σας, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στις Βρυξέλλες σήμερα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι η κυρία Ροζίτα Άγνιου, που είναι νομική μου σύμβουλος, που είναι υπεύθυνη για θέματα που έχουν να κάνουν ε, με τα άτομα με αναπηρίες, βρίσκεται μαζί σας. Μου ζητήσατε να θέσω το πλαίσιο, προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες σας και να βάλω κάποια προοπτική. Και θα το κάνω αυτό από την οπτική γωνία βέβαια του Ευρωπαίου Συνήγορου του Πολίτη. Ο Συνήγορο του πολίτη, να ξέρετε, ότι είναι το μόνο μη νομικό σώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει εντολή να εποπτεύει την συμμόρφωση των ευρωπαϊκών οργάνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα έτσι όπως αναφέρονται αυτά και για τα άτομα με αναπηρίες, όπως αναφέρονται λοιπόν μεταξύ άλλων στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ξέρετε, ο Ευρωπαίος ε, Συνήγορος του Πολίτη ασχολείται με τα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα, τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς και ερευνά τις καταγγελίες που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις τους. Ακούμε όλες τις καταγγελίες από όλες τις οργανώσεις και τα κινήματα, από όπου δηλαδή και αν μας έρχονται όσον αφορά τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες μεταξύ άλλων. Εμείς θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν φραγμοί, υπάρχουν εμπόδια ακόμα Ακούμε καταγγελίες από άτομα που λένε ότι έχουν δυσκολία πρόσβασης, για παράδειγμα στην ιστοσελίδα της ε, υπηρεσίας ε, επιλογής προσωπικού των ευρωπαϊκών οργάνων. Και εγώ το υπεθύμησα αυτό στην ΕΠΣΟ, ότι πρέπει να συμμορφώνεται με τη σύμβαση του ΟΗΕ και ότι πρέπει να λάβει υπόψη όλο όσα αναφέρει. Η ΕΠΣΟ μας ε, απάντησε θετικά προς αυτό. Έπειτα, τα άτομα που δουλεύουν για τα ευρωπαϊκά κοινωτικά όργανα επίσης έχουν επιστήσει την προσοχή μας σε αδυναμίες των ευρωπαϊκών κοινωτικών οργάνων όταν πρόκειται για παράδειγμα για τη φροντίδα των παιδιών τους με αναπηρίες ή ότι αποκλείονται τα παιδιά τους από τα ευρωπαϊκά σχολεία. Τώρα, άλλοι άτομα δηλαδή, πολίτες Ευρώπης που θέλουν να επισκεφθούν τα ευρωπαϊκά κοινωτικά όργανα, καταγγέλουν στον Ευρωπαίο Συνήγορο του Πολίτη ότι μερικές φορές δεν έχουν πρόσβαση στα κτίρια, ότι υπάρχουν προβλήματα και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή στην ιστοσελίδα ακόμα ε, των κοινοτικών οργάνων. Έτσι λοιπόν εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να δώσουμε λύσεις στις καταγγελίες αυτές. Εντοπίζουμε πρώτα απ' όλα τις αιτίε γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα γιατί υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν πλήρω στι συζητήσει, στις δράσει, στα προγράμματα και στι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά στα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μα ακριβώ αυτή είναι και η φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από τη σύμβαση του ΟΗΕ. Η ιδέα δηλαδή είναι ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίε είναι τελικά προβλήματα τη κοινωνία, και άρα εμεί πρέπει να φροντίσουμε να τα καταργήσουμε. Όπως ε, έχει εντοπίσει η πρώτη Ολομέλεια, πρέπει να την κάνουμε αυτή τη δουλειά, κυρίως τώρα σε περίοδο κρίσης. Και να φροντίσουμε, παρόλο που βρισκόμαστε υποποίηση να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει υποσχέσεις, υπογράφοντας και κυρώνοντας την ε, σύμβαση, Χωρί όμω να έχει αφιερώσει και του κατάλληλου πόρου. Όσον αφορά λοιπόν τη δικιά μου υπηρεσία, να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό όσον αφορά τον προπολογισμό του 2014, τη διαδικασία δηλαδή για τον προπολογισμό και βέβαια του, τη διαχείριση του προπολογισμού του 2013. Συγχρόνω, από δύο φορέ καταγγελίε που έχω πάρει, διαπιστώνω ότι μερικέ φορέ δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να κάνουμε το σωστό. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ε, έχω ασχοληθεί λιγάκι με το πιλωτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την κατάρτιση ατόμων ε, με αναπηρίες. Έχω πει λοιπόν ότι Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά και να μην τους αρνούμαστε ευκαιρίες εξαιτία της αναπηρίας τους. Το Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ε, σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους. Αυτό σημαίνει να μην δίνουν την εντύπωση ότι απασχολούν κάποιον επειδή είναι ανάπηρος και όχι επειδή είναι ικανός. Όχι, επειδή είναι ικανός καταρχήν ε, προσλαμβάνεται. Γιατί αν δεν το κάναμε αυτό, πλήττεται η ίδια η δημόσια εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ακριβώ έχω πει, σα τα παραθέτω. Και στην απάντηση που μου έδωσε το Κοινοβούλιο μου δίνει διάφορε λεπτομέρειε για τα βήματα που έχει αναλάβει προ τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα θα έρθω στην σύμβαση αυτή καθε αυτή. Στα πλαίσια τη εντολή του διαμεσολαβητή, του Ευρωπαίου Συνήγορου δηλαδή, οι πολίτε και διάφορες οργανώσεις στρέφονται προς εμένα εφόσον πιστεύουν ότι η δίκη τη ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δράσει σύμφωνα με τη σύμβαση. Εφόσον υπάρχουν τέτοιε λοιπόν καταγγελίες και φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα υπάρχουν όλο και περισσότερες, να ξέρετε ότι εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να στηρίξω τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες έτσι όπω αυτά εξασφαλίζονται από την σύμβαση. Ήδη από την αρχή ο συνήγορος του πολίτη πιστεύει ότι η εντολή του είναι ακριβώς ε, αυτή και αναφέρεται και στο άρθρο 33.2 πλαίσιο έτσι όπως αναφέρεται. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο Ευρωπαίος Συνήγορος είναι ένα από τα σώματα το οποίο έχει αναλάβει να προστατεύσει, να προωθήσει και να ελέγξει την ε, εφαρμογή της σύμβασης του ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας διαβεβαιώ ότι θα συμμετέχω στο πλαίσιο με πλήρη δέσμευση, γιατί θέλω να προχωρήσουμε με υψηλές φιλοδοξίες και να πάμε όσο γίνεται πιο μακριά όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη της σύμβασης. Προσβλέπω σε συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο. Ιδιαίτερα θέλω εδώ να αναφέρω την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία Έχω συνεργαστεί και κατά το παρελθόν και συνεχίζω να συνεργάζομαι στενά, όπω επίση και την Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει να παίξει ένα ρόλο κλειδί στηρίζοντα το έργο του πλαισίου μέσω του ελέγχου και των ε, ερευνητικών της δραστηριοτήτων. Τώρα για πόσας από εσά είναι εξοικειωμένοι με τη δουλειά του συνήγορου του πολίτη, γνωρίζετε ότι όταν δεσμεύονται απέναντι στους πολίτες τα κοινοτικά ευρωπαϊκά όργανα, κάνουν ό,τι μπορούν για να τα φέρουν και σε πέρας. Το ίδιο ισχύει και με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το ίδιο θα ισχύσει και με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Όσον αφορά εμένα, να ξέρετε ότι θα φροντίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις υποσχέσεις της απέναντι στους πολίτες βάσει της ε, σύμβασης που υπέγραψε και κύρωσε για τα άτομα λοιπόν με αναπηρίες. Ελπίζω αυτές οι παρατηρήσεις να σας βοηθήσουν στη συνέχιση του έργου σας και στις αποφάσεις που θα πάρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διαμαντούρο, για την παρέμβασή σας και με χαρά ακούμε από πλευρά σας την επιβεβαίωση ότι οι ίσες ευκαιρίες δεν κρίνονται με μέτρο το χρήμα, αλλά αποτελούν το μέτρο του Τη κοσμοθεωρίας μας, του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Θα παρακαλώσω λοιπόν τώρα τον κύριο Λάγκβατ, μέλος του EDF, να αναλάβει τον λόγο και να δώσει απαντήσεις στις παρατηρήσεις της κυρίας ε, Ματσόνη, τη κύρια Αντζελίλη, του κυρίου Διαμαντούρου. Έχετε το λόγο κύριε Λάγκβατ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα πρέπει να επιδείξουμε όλοι πλέον ευθύνη και να υλοποιήσουμε αυτά στα οποία έχουμε δεσμευθεί. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για την υλοποίηση της συμβάσεως για τα δικαιώματα και την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ και ξεκινώ από την ε, πραγματική κατάσταση που αντιμετωπίζω εγώ. Εγώ εξελέγην στην Επιτροπή με καθήκον, ως μέλος στην Επιτροπή, με καθήκον να παρακολουθούμε την υλοποίηση της συμβάσεως, της νομοθεσίας δηλαδή από τα κράτη-μέλη. Όταν λοιπόν συνέρχεται αυτή η Επιτροπή, καταγράφουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλούμε σε λογοδοσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τι έχει κάνει για να συμμορφωθεί με τις αρχές της συμβάσεως. Κάποια λοιπόν από τα ερωτήματα που έχουμε προς την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα εξής. Ερωτούμε λοιπόν πώς συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής, των πολιτικών επιλογών, οι ενώσει των ΑΜΕΑ, η οργάνωση των, οργανώση των πολιτών. Έχουν ληφθεί υπόψη οι εύστοχες παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή συνεργασία. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία σε τελευταία ανάλυση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Και πιστεύω ότι θα πρέπει η Επιτροπή να διατυπώσει το ερώτημα του τι μέτρα λαμβάνονται για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 33. Συγκεκριμένα, οργανωτικό πλαίσιο υπάρχει, έχει θεσπιστεί και αυτό που έχει θεσπιστεί θεωρείται ότι αρκεί για να δοθεί απάντηση στην πράξη για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν ε, οι ε, αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε ορισμένου τομεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σε κάποιου άλλου έχει μόνο συντρέχουσα αρμοδιότητα, ενώ σε κάποιου άλλου τομεί δεν έχει καθόλου αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτώ λοιπόν, είναι ανεξαρτήτως του που μένει ο, καθ... ο καθένας ε, για τον για το κάθε αμαία υπάρχει δυνατότητα να ξέρουμε ακριβώς τι είδους αρμοδιότητες υπάρχουν και υπάρχει πλαίσιο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε η πολιτική που εφαρμόζεται να έχει όντως ουσιαστικά αποτελέσματα για τα αμαία ανεξαρτήτως το που διαμένουν, τι είδους καθεστώς έχουν, σε ποια κατάσταση βρίσκονται γιατί νομίζω ότι στον τομέα αυτό χρειάζεται ακόμη περισσότερη πρόοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η Επιτροπή μα θέλει να ρωτήσει το εξής. Αυτό το οργανωτικό πλαίσιο είναι τόσο ανεξάρτητο και αυτόνομο όσο θα έπρεπε να είναι. διότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίζει ρόλο για την υλοποίηση της πολιτικής για τα ΑΜΕ, αλλά ταυτόχρονα έχει την ίδια, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εποπτεία του τρόπου με τον οποίο υλοποιούν τα κράτη-μέλη αυτή την πολιτική. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Ή μη τι άλλο μέχρι τώρα η Επιτροπή μας έχει μελετήσει το θέμα αυτό και της επιτήρησης ε, του μηχανισμού, δηλαδή το άρθρο 33 και θα, και θα θέλαμε να υπάρχει ένας αυτόνομος, ένας ανεξάρτητος μηχανισμός. Αυτό θέλουμε να επαληθεύσουμε. Από τις περιορισμένες γνώσεις που έχω όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη αυτό. Επίσης, ε, θα πρέπει να επαληθεύσουμε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοποίησης, φερειπίνη στην διεθνή συνεργασία σε σχέση με το άρθρο 32, μας απασχολεί το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαθέτει αναπτυξιακή βοήθεια κατά τρόπον ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και τα ΑΜΕΑ, στα κράτη τα οποία είναι, ε, υποφελούνται της αναπτυξιακής βοήθειας. Είτε πρόκειται για την Αφρική, είτε για τη Λατινική Αμερική, την ε, Νότια Αμερική Οπουδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει αναπτυξιακή βοήθεια, φροντίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς, ώστε να γίνεται το λεγόμενο mainstreaming, δηλαδή ενσωμάτωση των πολιτικών για τα αμαία σε κάθε τομέα δραστηριοποίηση μέσα από την αναπτυξιακή πολιτική και επίσης τα δικαιώματα που έχει εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι είναι επαρκή για να προωθήσουν ε, και να προαγάγουν μέσα στις κοινωνίες τα αμαία Εμείς αυτό θα το επαληθέσουμε πολύ επικριτικό πλεύμα. Επίσης, άλλη ερώτηση. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί τα μέσα του Διορθωτικού Ταμείου. Διότι μας φαίνεται παράδοξο μέσα κονδύλια του Ιδρυτικού Ταμείου να αξιοποιούνται για την ε, κατάργηση κάποιων θεσμών, θεσμικών οργάνων και την ε, θέσπιση κάποιων άλλων, όπως έχουμε δει σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως φέρει στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία κάναμε την τελευταία μας επαλήθευση, τη τελευταία συνεδρίαση σχετικά με την Ουγγαρία και διαπιστώσαμε αυτό το παράδοξο. Επίσης ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να επαληθευθεί είναι αυτό των πνευματικών δικαιωμάτων και των πιέσεων που ασκούνται στο επίπεδο αυτό. Στη διεθνή συνεργασία. ώστε και στην Διεθνή Οργάνωση για τα Πνευματικά Δικαιώματα να εξασφαλίζονται μέτρα για την πρόσβαση σε πνευματικό προϊόν, βιβλία και ούτω καθεξής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πώς θα αυτή η πρόσβαση σε βιβλία. Πώς θα μπορούμε να ξέρουμε τι είδου ε, δυνατότητες έχουμε και ότι μπορούμε να διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο με αυτό που διάβασε και η φίλη εδώ, η Μάργαρετ Άουκεν, η Δανή Ευρωβουλευτής. Πρέπει νομίζω πάντοτε να έχουμε το βλέμμα στραμμένο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κοιτάμε ότι πράγματι εφαρμόζονται σωστά οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, να δίνονται απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βλέπουμε τις εκθέσεις και κυρίως να δούμε και την έκθεση βέβαια της Επιτροπής μας το 2013. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Στέιγκ, μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε την Ολομέλεια. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην Ολομέλεια, θα ήθελα να ζητήσω από τον Κίκο Γκέντς, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπρόεδρο της Διακομματικής Ομάδας για τα άτομα με αναπηρία και Γενικός Γραμματέας του EDF, να προεδρεύσει το επόμενο μέρος της Συνόδου. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ευχόμαστε ότι θα παραμείνετε και πιστοί στο χρονοδιάγραμμα. Είναι εδώ που Good morning. Ε, good morning. Καλημέρα σας. Πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο μας. Γι' αυτό θα σας ζητήσω να ξεκινήσουμε με αυτή τη δεύτερη περίοδο της σημερινής μας συνάντησης ευθύς αμέσως. Σας καλωσορίζω και εγώ όλους εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Βαδακαστάνου με τον οποίο από κοινού προεδρεύουμε. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να τηρηθεί ο χρόνος και ελπίζουμε πως όλοι αυτοί που έχω στον κατάλογο μιλητών θα έχουν αρκετό χρόνο για να παρέμβουν. Θα σας πω λίγα εισαγωγικά μόνο σχόλια. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι μια πολύ δυνατή στιγμή αυτή για όλους εμάς που εκπροσωπούμε διάφορες οργανώσεις από διάφορες χώρες. Αλλά ακόμα περισσότερο πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μας που είμαστε ευρωβουλευτές και βλέπω στην αίθουσα πολλούς. Για όλους εμάς λοιπόν που έχουμε έτσι την ευκαιρία να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τα σχόλιά σας, και να σας ε, καλωσορίσουμε εδώ στην, ε, στο χώρο μας να μάθουμε από σας και να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος να μάθουμε από σας και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις ε, μαζί. Σίγουρα Το ξέρουμε όλοι ότι σε περίοδους κρίσης η ζωή γίνεται πιο δύσκολη για όλους. Ακόμα περισσότερο όμως για εκείνους που ζουν με κάποιες δυσκολίες, με κάποιες αναπηρίες. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να λαβαίνουμε υπόψη μας τις δυσκολίες αυτές. Η κρίση εξάλλου δεν είναι μόνο μια οικονομική, μια δημοσιονομική κρίση. Βλέπουμε ότι είναι μια κρίση γενικότερη που περιορίζει τις δαπάνες για την απασχόληση, για την εκπαίδευση, για τις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν επιτυχάνεται έτσι η ισότητα στην Ευρώπη. Είναι και μια κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλές χώρες. Γι' αυτό και πρέπει να συνεργαστούμε, να κάνουμε βήματα προς τα μπρος για να τα καταφέρουμε. Έχω πέντε λεφτά στη διάθεσή μου, οπότε δεν θα μακρηγορήσω. Απλώς να πω ότι αυτή την εποχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε το πλαίσιο για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Κάτι το οποίο θα είναι αποφασιστική σημασίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών. Ακούσατε ήδη τις δυσκολίες ότι γίνονται δράστιες συζητήσει και μεταξύ των χωρών μελών αλλά και μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Σας διαβεβαιώ ότι οι Ευρωβουλευτές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά στηρίζει όλες τις φιλοδοξίες που έχουμε κι εμείς εδώ διατυπώσει. Εγώ προσωπικά είμαι εισηγήτρια για το πρόγραμμα όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, οπότε θέλω να φροντίσω οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματά τους για να μπορούν να τα ασκούν και καλύτερα και βέβαια να προστατεύονται σε όλες τις χώρες μέλη. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για το ταμείο αυτό και προσπαθούμε και εμείς να συμπεριλάβουμε και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Δεν είμαστε στο τέλος των διαπραγματεύσεων ακόμα με το Συμβούλιο, πάντως συζητάμε και στη βάση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες στη ρύθμιση αυτή. Θέλουμε να μιλήσουμε για την προσβασιμότητα, για την ε, εφαρμογή της σύμβασης από τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε όλες αυτές οι πτυχές να παραμείνουν μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων και ότι θα μπορέσουμε τα κονδύλια αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε και τα επόμενα 7 χρόνια. Γνωρίζετε ότι και η νομοθετική πτυχή είναι πολύ σημαντική και η εφαρμογή είναι πολύ σημαντική, αλλά βέβαια και οικονομικοί πόροι προκειμένου να γίνει η εφαρμογή αυτή και να πετύχουν οι φιλοδοξίες μας και στόχοι μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάλι που είστε εδώ και ο κύριος Κατάνη τώρα θα πάρει το λόγο για να μιλήσει στο σώμα. Και μετά όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ και που θέλετε να παρέμβετε θα μπορέσετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Κατάνη. Ο κύριος Ροντόλφο Κατάνη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, οι προλαλήσαντες είπαν πολλά σημαντικά για την ε, διάσκεψη, για τη σύμβαση των Εθνών. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε σήμερα, για μένα, είναι μάλλον να επιμείνουμε στις συνέπειες της κρίσης μιας κρίσης η οποία μετατρέπεται σιγά σιγά, μάλλον όλο και πιο πολύ, σε κρίση των ανθρωπινών δικαιωμάτων, να παράσει κρίση οικονομική ή δημοσιονομική. Τα μέτρα λιτότητας υπάρχει κίνδυνος να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια περιοχή φτωχή, οι συνθήκες διαβίωσης για τα αμαία είναι χειρότερες, τα κοινωνικά, τα κοινωνικά δικαιώματα κινδυνεύουν ως συνέπεια των περικοπών στα επιδόματα και, τις, ε, ε, και τη βοήθεια, την υποστήριξη. Ιδιαίτερα πλήττονται τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, καταργούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες και έτσι υπονομεύεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην, κοινωνία, στην ε, αλληλεγγύη και την κοινωνική ενσωμάτωση. Όπως είπα λοιπόν η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι πάνω απ' όλα κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. η ευρωπαϊκή θεσμοί, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αναζητήσουν το δρόμο διεξόδου από τον εφιάλτη αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με 24 από τα 27 κράτη-μέλη έχει κυρώσει ε, την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και έχει πλέον την υποχρέωση η Ένωση και τα κράτη-μέλη να την υλοποιήσουν. Και καθώς είναι συμβαλόμενο μέρος και η ίδια η Ένωση, έχει και εκείνη, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, την υποχρέωση για εφαρμογή της σύμβασης. Έτσι λοιπόν πρέπει να δημιουργήσει μια κοινωνία ε, ευρεία, βιώσιμη, αηφόρο δηλαδή με κοινωνική συμπερίληψη και για τα άτομα με αναπηρίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως ακόμη να το έχει επιτύχει αυτό, δεν έχει καν πλησιάσει στους στόχους, ούτε καν στρατηγίες του 2020. Άρα λοιπόν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει ένα ισχυρό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ένα σύνολο μέτρων και κοινωνικές επενδύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, θα επενδύσει σε κοινωνικέ πολιτικές και υπηρεσίε που θα συμβάλλουν στην δημιουργία μια πιο, ε, μια πιο ανοιχτής, μιας πιο ανοιχτής, μιας πιο ευημερούσας, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Ένα πακέτο λοιπόν, μια δέσμη κοινωνικών μέτρων που θα πρέπει να σημαίνουν την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ με κατάλληλους πόρους και κοινωνική προστασία για την συμμετοχή στην αγορά εργασίας και για αντιστάθμιση όπου υπάρχει απουσία εισοδήματος από εργασία αλλά και αποδεκτή πρόσβαση, ικανοποιητική σε οικονομικούς όρους πρόσβαση και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της υπηρεσίας υγείας. Πρέπει λοιπόν τα ΑΜΕΑ να βρουν τη θέση τους και σαν καταναλωτές μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά. Το EDF ε έχει κάνει σαν κύρια εκστρατεία για το 2012 τρία βασικά ζητήματα, την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, των υπηρεσιών και των αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την υιοθέτηση ενός, μιας ευρωπαϊκής πράξης, νομοθετικής πράξης προσβασιμότητας και το ζήτημα της οδηγίας για την προσβασιμότητα των δημοσίων ε, ιστοτόπων και ιστοτόπων παρέχουν ε, υπηρεσίες στο ευρύ κοινό. Προσβασιμότητα λοιπόν που πρέπει να είναι η κύρια, η κατευθυντήρια γραμμή και στο διάλογο για, και στις διαδικασίες για τις δημόσιες προμήθειες και στις παροχές από τις δημόσιες αρχές. Χρειάζεται και ακούστηκε και νωρίτερα να υπάρχει τόσο το δημοσιονομικό όσο και το πολιτικό πλαίσιο αλλά σε όρους ισχυρούς και στεναρούς και είμαστε ακόμη σε μια προσπάθεια και ενώ είμαστε ακόμη σε μια προσπάθεια, σε μια απόπειρα περικοπής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, εμείς ζητούμε τουλάχιστον 25% του Ταμείου Συνοχής να αφιερώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Προπολογισμό να υποστηρίζει τι κοινωνικέ υποδομέ, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, να μειώνει τι ανισότητε και την φτώχεια, ενώ οι περικοπέ στι κοινωνικέ δαπάνε γεννούν ενεργεία και η υποβάθμιση τη κοινωνική κατάσταση και αντίστοιχα οι ε, ανησυχητικές πολιτικές εντάσεις. Αυτή τη στιγμή η φτώχεια αυξάνεται, δεν μειώνεται Αντί για κοινωνική συνοχή αντιμετωπίζουμε ανισότητες, αποκλεισμό, διακρίσεις και αναμένουμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναλάβουν δράση με κύριο γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, ιδάλλως θα απολέσουν την αξιοπιστία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, υπάρχουν σημαντικές προσδοκίες από πλευρά των ΑΜΕΑ, τόσο για τη δράση μέσα στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να ε, υλοποιήσουν αυτές, να κάνουν πράξη αυτές τις προσδοκίες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ κύριε Κατάνη για την ε, παρέμφαση σας. Από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους, δύο εκ των συναδέλφων ευρωβουλευτών, συναδελφοί, που δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγο νωρίτερα στο προηγούμενο κομμάτι της συστήσεως, η κυρία Γκάμπρι Τσίμερ της ε, Γκουε, πρόεδρος της ομάδας της ε, ΓΚΟΕ, και ο κύριος Ρουέδα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος των Πρασίνων, έχουν ζητήσει να παρέμβουν τώρα. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε με εσά και μετά να συνεχίσουμε με τους λοιπούς ομιλητές. Γκάμπι, παρακαλώ, πώς να λάβεις το λόγο. Ευχαριστώ θερμά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω σήμερα σε αυτό το κοινοβούλιο των ατόμων με ειδικέ ανάγκε Εντυπωσιάζομαι, πρέπει να σα πω βαθιά, από τα όσα άκουσα και είδα σήμερα διότι τα προβλήματα των ΑΜΕΑ διαπιστώνω ότι δεν είναι προβλήματα μιας ιδιαίτερης χωριστής ομάδας ανθρώπων που έχουν αναπηρίες. Είναι προβλήματα τα οποία μας αφορούν όλους. Είναι προβλήματα της καθημερινής ζωής που εθίγησαν σήμερα και που πρέπει από κοινού να επιλύσουμε όλοι. Γι' αυτό είμαι υπερήφανη που έχω την ευκαιρία εδώ να σας καλωσορίσω όλες και όλους και που μπορώ να συμμετάσχω σε αυτόν τον κοινό διάλογο μαζί σας. Ένα διάλογο μεταξύ εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρίες, των πολιτικών εκπροσώπων ε, των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλουμε ασφαλώς να ενισχύσουμε. Ελήψη χρόνου θα, θα προσπαθήσω να περιορίσω την παρέμβασή μου στο ελάχιστο. Άκουσα πολύ ενδιαφέρουσε παρατηρήσεις από τους ομιλητές εδώ στο Προεδρείο ότι πρέπει να κοιτάξουμε την στάση των ευρωπαϊκών οργανών και ιδιαίτερως πρέπει να ασχοληθούμε με τον τρόπο με τον οποίο η αναπτυξιακή βοήθεια ιδιαίτερως μπορεί να συμβάλλει περισσότερο και καλύτερα στην προστασία και τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και στα φτωχότερα κράτη του κόσμου. Ιδιαίτερα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να σας πω εμείς ε, και με τις αντιπροσωπείες μας, ε, αντιπροσωπεία παραδείγματι για τις σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ, Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού, έχουμε επεξεργαστεί έκθεση για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίε και θεωρώ ότι η έκθεση αυτή έχει πολύ μεγάλη και ζωτική σημασία γιατί καθιστά σαφέστατο ότι στη δουλειά μας για μας του ίδιους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε τους περιορισμούς και να υποστηρίξουμε ιδιαίτερω τα μέσα, ε, τα προγράμματα εκείνα με ιδιαίτερου πόρους που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα μέσα για τα άτομα με αναπηρία, που μπορούν δηλαδή να τα στηρίξουν στην καθημερινή του ζωή. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφέρω ε, μια άλλη παρατήρηση πριν ε, να γίνω ευρωβουλευτή, ε, που δούλευα στο κρατήδιο τη Τουρκία στη Γερμανία, είχα πολλέ επαφέ ε, στην επαγγελματική μου, στον επαγγελματικό μου βίο με γυναίκε ιδιαίτερω που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρία και κυρίω το πρόβλημα, με είχε απασχολήσει το πρόβλημα τη βία εις γυναικών με αναπηρίε. Και πιστεύω ότι σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε τι ε, συζητήσει μα σε κάποιο χρονικό σημείο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα στι πραγματικέ του διαστάσει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ε, μπορούν οι αρχές, οι επίσημες αρχές να στηρίξουν, να βοηθήσουν τις γυναίκες αυτές, να τις προστατέψουν, τις γυναίκες με αναπηρίες από τη βία Και ε, μια τρίτη παρατήρηση, επίση πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι ναι, βρισκόμαστε εν μέσω κρίση, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται βέβαια για μια πολύ βαθιά κρίση. Και πιστεύω ότι ε, από κοινού αυτό που θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να εμποδίσουμε μία εξέλιξη κατά την οποία η δημοσιονομικές εξελίξεις θα είχαν σαν συνέπεια, δηλαδή η κατάρτιση των προϋπολογισμών θα έχει σαν συνέπεια να αποκλείονται τα αμαία από την κοινωνία στην οποία ζουν, να μην μπορούν δηλαδή να βρίσκουν πρόσβαση είτε στη δημόσια υπηρεσία είτε στην, ε, στην αντιμετώπιση, στην επίλυση των προβλημάτων που βιώνουν και νομίζω ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καθήκον να το επιδιώξει, αλλά και το σημερινό, το δικό σας Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο των ΑΜΕΑ, πρέπει να έχει τη δυνατότητα της πρόσβασης στη δημόσια υπηρεσία, στο δημόσιο αγαθό και να απαιτήσουμε ο δημόσιος χώρος να επανέλθει μέσα στην κοινωνία και να ξαναεγγραφεί μέσα στην κοινωνία μας, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την τάση για ιδιωτικοποιήσεις η οποία ουσιαστικά περιορίζει και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας. Αυτό λοιπόν είναι το ε, κύριο αίτημα, η κύρια παρατήρηση που είχα να κάνω με αυτή τη σύντομη παρέμβαση. ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνεργασία σας, στην τωρινή και την περαιτέρω και ιδιαίτερο στην υλοποίηση της, Ευρω... της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, για την οποία από κοινού αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ραούλ Ρομέρα Ιρουέδα, αντιπρόεδρο των Πρασίνων. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ήθελα να είμαι βέβαιος γιατί παρακολουθώ προσεκτικά τις συζητήσεις μέχρι τώρα και πρέπει να πω ότι όλα αυτά είναι ακριβώς αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως μέλος των Πρασίνων. Εμείς αυτή την εβδομάδα εστιάσαμε τις εργασίες μας σε πολλούς τομείς. Αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα από τα θέματα που κατά την απόψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για το ζήτημα της ε, οριζόντιας οδηγίας ε, κατάργησης των διακρίσεων που βρίσκεται τώρα στο Συμβούλιο. Εγώ είμαι συγκεκριτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Οι δυσκολίες που βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια έχουν να κάνουν με την κακή αντίληψη ενός ε, προβλήματος ε, του κόστους της αντίληψης που έχουν ορισμένα κράτη-μέλη ότι είναι υπερβολικά ακριβή η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Άκουσα προσεκτικά τα όσα είπατε πολλοί από εσάς σήμερα το πρωί και πιθανώς ε, θα συνεχίσετε να τα λέτε περισσότεροι. Αυτά ακριβώς είναι αυτά που πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι. Να ε, υπερασπιστούμε ενώπιον ορισμένων κρατών που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επένδυση σε θέματα συνοχής είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παραλείψουμε σε περίοδους κρίσης. Αυτό είναι το λάθος το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη φάση της ιστορίας μας. Ελπίζω, όπως υπόθηκε και το επικυρώνω και εγώ, ότι η υπογραφή της συνθήκης ε, των ΗΠΑ για τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να αποτελέσει τρόπο ενίσχυσης των νομικών υποχρεώσεων επέκταση της προστασίας κατά των διακρίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως βάση για να πείσουμε όλα τα κράτη-μέλη και ειδικότερα εκείνα τα οποία ακόμα αναρωτιούνται κατά πόσο είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η επέκταση της ε, αρχής της μη διάκρισης ε, σε ολόκληρη τη νομική σφαίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες, γιατί εδώ μιλάμε για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν να βλέπουν να εκπληρώνουν τα δικαιώματά τους, να διασφαλίζονται και να εξασφαλίζονται οι ίσες ευκαιρίες ε, που πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα άτομα ανεξαρτήτως της κατάστασής τους. Αυτή η εκδήλωση πιστεύω θα μπορέσει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς ορισμένα κράτη-μέλη εξακολουθούν να προσπαθούν να αποκρύψουν την αντίθεση τους ε, πίσω από πολύ σαθρά επιχειρήματα κόστους δαπανών της πρότασης ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα επιχειρήματα ε, ζητήσαμε να γίνει μια μελέτη για να αναδείξουμε όχι μόνο τα κόστη αλλά και τα ωφέλη της συνοχής καθώς και τα ωφέλη τα κοινωνικά, όχι μόνο τα ατομικά τα ωφέλη που προκύπτουν από, αυτούς, από την εφαρμογή αυτών των νόμων κατά των διακρίσεων. Ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή διστάζουν να υιοθετήσουν αυτά τα πρότυπα θα καταλάβουν κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τα υιοθετήσουν στο, η μεγάλη πλειοψηφία των ομάδων στο Κοινοβούλιο το υποστηρίζει και σας παροτρύνω και με βέβαιος ότι το ψήφισμα που και την περασμένη εβδομάδα στο Συμβουλίο βάσει του άρθρου 265 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε έγκριση της οδηγίας το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, ε, ουσιαστικά μιλάμε για ένα ζήτημα δικαιωμάτων. Προσβασιμότητα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με δημόσια και τα κοινά. Σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε στην ομάδα των Πρασίνων ε, ουσιαστικά ε, το θέμα της δημοκρατίας σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη με μια νέα ερμηνεία που χρησιμοποιείται στη δική μας ομάδα με την διερμηνία ομιλίας σε κείμενο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένας φυσιολογικός τρόπος πρόθεσης της δημοκρατίας σε όλες μας τις συζητήσεις, ακόμη και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι το θέμα της εκδήλωσης αυτής δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση, αλλά κανόνας. Κάτι το οποίο θα προωθείται φυσιολογικά, ανεξαρτήτως κόστους, διότι επιμείνω. Δεν είναι μόνο θέμα δαπανών που ορισμένοι χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία, αλλά είναι θέμα ουσιαστικά ωφελών. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που εδώ το συζητάμε αυτό και χαρακτηρίζει πολλές από τις συζητήσεις μας. Και χαίρομαι που η μεγάλη πλειοψηφία των ομάδων ε, υποστηρίζει αυτό το όρομα, αυτή την αντίληψη. Ο μόνος τρόπος ουσιαστικά να καταλάβουμε αυτή την πρόπτικη αυτό το πρίσμα των ίσων ευκαιριών. Ε, Ευχαριστούμε πολύ αν δεν σας πειράζει, κάποιοι από τους συναδέρφους μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να φύγουν. Η Λίζαπετ, για παράδειγμα, έχει ζητήσει το λόγο αν μπορείς κάπως ε, σύντομα τώρα, γιατί ξέρω ότι μετά πρέπει να αποχωρήσεις. Από τους πράσινους, ε, λοιπόν, η Λίζαπετ Σλάκη. Κύριε Σρότερ, Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Θα μιλήσω κι εγώ τη μητρική μου γλώσσα. Ελπίζω ότι θα με παρακολουθήσετε και με τα ακουστικά. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μιας επιτροπής δηλαδή η οποία χειρίζεται πολλά θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν ευθέως τα ΑΜΕΑ, μια επιτροπή η οποία είναι στρατευμένη στον αγώνα αυτό και πρέπει να πω ξεκινώντα ότι έχουμε εκπονήσει έκθεση για την στρατηγική τη σχετική με τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον συνάδελφο Άνταμ Κόσα που κάθεται ακριβώ δίπλα μου και έχουμε ε, επιτύχει πιστεύω ε, με συνεργασία μεταξύ μας μια πολύ καλή έκθεση μια έκθεση όπου μπορούμε στα λεγόμενα ήπια μέτρα πολιτικής να εξασφαλίσουμε ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή πολιτική. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι παρατηρείται με πολύ μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο της διαγραφής της ε, αρρωγής που προσφερόταν μέχρι τώρα στα ΑΜΕΑ στην Ελλάδα και ότι φοβόμαστε ότι επιδεινώνεται ριζικά η κατάσταση για, την, ε, για το, τα ΑΜΕΑ στην Ελλάδα, μια κατάσταση στην οποία δεν αποδεχόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε επικρίνει μαζικά την Τρόικα για τις επιλογές της αυτές. Ε, επίσης θα ήθελα να επισημάνω στην Επιτροπή Απασχόλησης έχουμε προβλέψει την εκπόνηση μιας ε, εκθέσεως πρωτοβουλίας για την υλοποίηση της οδηγίας κατά των διακρίσεων ως προς την πρόσβαση στον χώρο εργασίας και την απασχόληση ε, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να θέσουμε το δάκτυλο επί το τύπο των Ήλων και να καταγράψουμε την πραγματικότητα στην Ευρώπη όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας κατά των διακρίσεων. Δηλαδή την απέτηση για μια ελεύθερη και χωρίς ε, προσκόμματα προσβάσεως στην κατάρτιση, στην απασχόληση για τα άτομα με ε, αναπηρίες. Χωρίς να εμποδίζονται αυτά λόγω της αναπηρίας τους από την πρόσβαση. Επίσης, σημειώνουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές, ε, πάρα πολλές πραγματικά εκδηλώσεις και ε, συνεδριάσεις, ειδικότερα για το Διαρθρωτικό Ταμείο, αλλά και για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και θέλουμε το, ε, τα Διαρθρωτικά Ταμεία να υλοποιούνται κατά τρόπον ώστε να καταργούν τα εμπόδια να παραμερίζουν τα προσκόμματα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε τα διαρθρωτικά ταμεία να είναι διαρθρωμένα έτσι ώστε να συμμετέχουν σε αυτά και τα ΜΕΑ στο σχεδιασμό τους. Και ιδιαίτερα θα αναφερθώ πάλι στον Άνταμ Κώσα, ο οποίος είναι ε, και μέλος της Επιτροπής ε, διαπραγμάτευση. Μάλλον προσπαθούμε να, τον να του εξασφαλίσουμε θέση στην Επιτροπή Διαπραγμάτευση. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, αλλά άνταμ θα τα καταφέρουμε, σε διαβεβαιώ. Και θα ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο, μια και είμαι από τη Γερμανία. Ε, να πω λοιπόν ότι με πολύ μεγάλη ανησυχία βλέπω το γεγονός πως η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιτάσσεται στην πέμπτη οδηγία για, διακρί, για τις διακρίσεις, για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι υπάρχουν ε, κρατήδια στη Γερμανία τα οποία μεριμνούν ως προς την ε, ε, εξέλιξη των ανοιχτών λεγόμενων σχολείων ή σχολείων κοινωνικής ενσωμάτωσης στο εσωτερικό τους και δεν έχει κανένα πλέον επιχείρημα βάσιμο η γερμανική κυβέρνηση, η ομοσπονδιακή δηλαδή κυβέρνηση, ώστε να παρεμποδίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την έγκριση αυτής της πέμπτης οδηγίας κατά των διακρίσεων. Θέλουμε λοιπόν να σταματήσει αυτή η αντίδραση, αυτό το βέτο και να προχωρήσουμε εντατικά προς την πρόοδο για την πέμπτη οδηγία κατά των διακρίσεων, ώστε να αλλάξει η γερμανική κυβέρνηση τη στάση τη για το θέμα αυτό, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να θεσπίσουμε δίκαιο και μάλιστα ατομικά δικαιώματα για τα αμαία ω προ την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση. Αυτό είναι ο στόχο μα. γι' αυτό αγωνιζόμαστε και στην τρέχουσα θετία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε θα τα καταφέρουμε. Σα ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σρέτερ, κύριε Σεκουτάνη. Πράγματι, οδηγία για την κατάργηση των ε, διακρίσεων σε κάποιο σερτάρι έχει χωθεί. Από το 2008 δηλαδή κοιμάται. Νομίζω ότι πρέπει να ξυπνήσει, όπως είπατε κι εσείς. Πρέπει να αγωνιστούμε για την κατάργηση των διακρίσεων και να μην επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να δυσκολεύουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Τώρα, συνεχίζουμε και πάμε στις παρεμβάσεις των εκπροσώπων μας που έχουμε εδώ, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Αυτό Κοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρίες. Έχετε δύο λεπτά ο καθένας στη διάθεσή σας και θα ήθελα να αρχίσω με την κυρία Μαλία Γκρίνερ, Αυστρία, από το Εθνικό Συμβούλιο της Αυστρίας για άτομα με αναπηρίες. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ απαιτώ να μην υπάρχουν να μην υπάρχουν εμπόδια ή προσκόμματα σε οδήποτε επίπεδο, είτε σε επίπεδο σωματικών εμποδίων, φυσικών εμποδίων, ηθικών εμποδίων και απαιτώ να υπάρχει ε, η δυνατότητα σε κάθε επίπεδο της σχολικής ε, πορείας ενός παιδιού αυτή η απαλλαγή από εμπόρια, από εμπόδια, από φραγμούς ώστε να μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση όπως κάθε άλλο παιδί, το, το παιδί με ειδικέ με αναπηρίες αλλά και ο επαγγελματίας στην πρόσβαση στην εργασία και ο δάσκαλος ή η δασκάλα με αναπηρίες και να προσφέρεται επαρκής υποστήριξη στα παιδιά με ε, ιδιαίτερες ανάγκες μαθησιακές και ε, να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, για να οποιοδήποτε θέλει, θέλει να ε, εξειδικεύσει στον τομέα αυτόν. Ε, I am, I am... με χαρά Βλέπω ότι είναι πολλοί οι ευρωβουλευτές εδώ παρόντες. Ε, κάποιοι όμως ίσω χρειαστεί να αναποχωρήσουν κάποια στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνήσαμε με τον κύριο Κατάνη να ακούμε μία παρέμβαση από τις εθνικές ε, αντιπροσωπείες και μία από τους ευρωβουλευτές, ώστε να δοθήσουμε αρκετό χρόνο για όλους. Παρακαλώ λοιπόν την κυρία Λοπέ Φοντανιέλ να λάβει το λόγο. Παρακαλώ όμω αυστηρά δύο λεπτά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να ακούσουμε και τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Λίγα έχω να πω. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Εγώ προέρχομαι από το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και συμμετέχω στην Επιτροπή Απασχόλησης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές λοιπόν για τα θέματα τα κοινωνικά και κυρίως για το θέμα των ε, αναπήρων συμφωνούμε. Συμμερίζομαι λοιπόν απόλυτα τα όσα είπε η κυρία Κόνς πριν, όπως επίσης και η συνάδελφος Σέντερ και δεν θα τα επαναλάβω. Πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Εδώ ήρθαμε για να ακούσουμε. Υπάρχει ένα σημαντικότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και αυτό είναι και το κύριο σε όλες τις χώρες και στη δικιά μου πολύ περισσότερο, που είναι η ανεργία. Δυστυχώς τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερες δυσκολίες για να έχουν πρόσβαση στην εργασία, χάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους και έχουν λιγότερες δυνατότητες κατάρτισης. Η λιτότητα δυστυχώς είναι μια αναγκαιότητα και στην Ισπανία, αλλά πρέπει να φροντίσουμε η λιτότητα αυτή να μην πλήττει περισσότερο ε, τα άτομα που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε, πιστεύω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ε, η επόμενη ομιλήτρια μάλλον, είναι η κυρία Πασκάλα Ρίμπ ο κύριος Πασκάλερ, η κυρία Ρίμπα από το Γαλλικό Συμβουλίο για άτομα με αναπηρία. Θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα και τις ελλείψεις μετά από την θέση σε ισχύ της συνθήκης ε, το Μάρτιο του 2010 στη Γαλλία. Για τη Γαλλία πρόκειται για ένα μείζον πολιτικό εργαλείο, ένας πραγματικός μοχλός ε, για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία θα έλεγα ότι έχουμε την κατάσταση πριν και μετά την κύρωση της συνθήκης. Τα αποτελέσματα μετά από τη θέση ισχύ της συνθήκης θα έλεγα ότι αυτή η συνθήκη έδωσε στη γαλλική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία μια νέα πνοή και μεγάλη δύναμη στο κίνημά μας για την υπεράσπιση των ατόμων βασιζόμενη στα δικαιώματα και όχι ε, σε ε, καλές πράξεις. Ε, μας βοηθάει να πάμε πολύ πιο πέρα από την απλή νομοθεσία που είχαμε μέχρι τότε προκαλεί αλλαγές ε, στην εκπόνηση πολιτικών. Δεν μιλάμε πια για ατομικέ πολιτικές προσαρμογής, αλλά στο σχεδιασμό μιας κοινωνίας ανοιχτή για όλους. Πιο συγκεκριμένα είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση τον περασμένο Σεπτέμβριο μια συγκυκλίου του Πρωθυπουργού σε σχέση με τη συνεκτίμηση των αναπηριών σε όλα τα νομοσχέδια υπέρ μια οριζόντιας πολιτικής. Για πρώτη φορά έχουμε ένα επίσημο γαλλικό κείμενο του Πρωθυπουργού που βασίζεται στη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών και που επιβεβαιώνει ότι πρέπει να αποτελεί το εφαλτήριο για συγκεκριμένες διατάξεις για άτομα με αναπηρία σε όλα τα μελλοντικά νομοσχέδια. Επίσης έχουμε ένα διαγνωστικό δελτίο για τα άτομα με αναπηρία που θα συνοδεύει, θα επισυνάπτει σε όλα τα νομοσχέδια στο εξή. Όσον αφορά τι ελλείψει μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη, θα έλεγα ότι σήμερα ε, παρατηρούνται πολλές αποκλήσεις ε, ε, μεταξύ γαλλικής νομοθεσίας και της Σύνθηκης των Ηνωμένων Εθνών. Στη γαλλική νομοθεσία διατηρείται η ιατρική πτυχή χωρίς να μιλάμε για την παιδεία χωρίς διακρίσεις, την αυτονομία διαβίωσης και τη νομική προστασία. Η Γαλλία λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσει τη νομοθεσία τη, ώστε να συμμορφώνεται αυτή με τη συνθήκη των Εθνών. Θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδη ελευθερίες δεν μπορούν να ε, ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες. είμαστε εντελώς ίσοι ή όχι. Και όπως είχε πει ο Γκάντι, κάθε συμβιβασμός βασίζεται σε παραχωρήσεις από όλα τα μέρη. Δεν μπορούν να υπάρχουν όμως αμοιβέ παραχωρήσει όταν μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την κυρία Σιλβάνα Ράπτη, τη συναδελφό μου, Ευρωβουλευτή, να λάβει το λόγο για δύο λεπτά. Έχετε δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ Είμαι ε, στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι αισθάνομαι χαρά, αισθάνομαι τιμή, αλλά ταυτοχρόνως αισθάνομαι και μεγάλη ευθύνη που βρίσκομαι εδώ στο Τρίτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία. Η σημερινή συνάντηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα της είναι εξαιρετικά σημαντικό και ουσιαστικά και ουσιαστικό η εφαρμογή της σύμβασης του οηε για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι η αρχή της μη διάκρισης η αρχή της αποδοχής της διαφορετικότητας του κάθε ατόμου η αρχή της ισότητας των ευκαιριών ενώ πρέπει να θεωρούνται αυτονόητες σε κάθε προηγμένη κοινωνία βλέπουμε στην πράξη ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο πάνω σε αυτή την κατάσταση έρχεται να προσθεθεί η οικονομική κρίση την οποία οικονομική κρίση δέχονται στους ώμους τους περισσότερο δύσκολα περισσότερο βαριά από κάθε άλλον τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους. αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το επιτρέπουμε τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να εξαιρούνται από τα πακέτα λιτότητας τα οποία εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες ανάμεσά τους και η ελλάδα που βρίσκονται σε πρόγραμμα. διαφορετικά κινδυνεύει ο κοινωνικός χαρακτήρας της ευρώπης. θεωρώ ότι πριν απ' όλα εμείς οι ευρωβουλευτές εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα δράσης όπως και οι συνάδελφοί μου ανέφεραν στην καθημερινή μας δουλειά νομοθετώντας και προσθέτω και τη δική μου μικρή συμβολή τη δική μου μικρή προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση. έχω καταθέσει γραπτή ερώτηση στην κομισιόν με την οποία ζητώ να πληροφορηθώ τι σκοπεύει να κάνει η κομισιόν ώστε να, μπορεί να, παρακολουθούν, να μπορούν να παρακολουθούν τα άτομα με ακουστικά προβλήματα όλες τις συνεδριάσεις και τις εργασίες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τους θέλουμε όλους εδώ να μπορούν να παρακολουθούν, να συμμετέχουν και να παρεμβαίνουν στη δουλειά μας για να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς. Ευχαριστώ. Yeah, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ράπτη. Επόμενος ομιλητής από τη Δανία, ο κύριος Τόλκιν Όλεσεν, από τον Οργανισμό Ατόμων με Αναπηρία της Δανίας. Τόλκιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια για τη συνθήκη στην οποία αναφερθήκαμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις τεράστιες προσπάθειες που έχει κάνει για να πείσει την Κομισιόν να μην αντιτεθεί πλήρως ε, στη συνθήκη, ουσιαστικά να την υποστηρίξει ώστε να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα όρασης και ανάγνωσης ε, από το να έχουν πρόσβαση σε κείμενα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι τα άτομα με προβλήματα όρασης και δυσκολίες ανάγνωσης θα μπορούν έτσι να έχουν πρόσβαση σε βιβλία. Δεν έχουμε πρόσβαση σε βιβλία. Δεν μεταφράζονται. Αν μεταφραστούν θα μπορούμε να έχουμε πλήρη πρόσβαση στην κοινωνία. Θέλουμε έτσι πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην παιδεία και στην απασχόληση. Χωρίς αυτή την πρόσβαση δεν μπορούμε να συμβάλλουμε στην κοινωνία όπως θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε επίσης να εξελιχθούμε σε εξαιρετικούς καταναλωτές. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή κοινότητα να ξεφύγει από αυτή την κρίση. Θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στο σύνολο της κοινωνίας, να ενισχύουμε την κοινωνία, να συμβάλλουμε οικονομικά. Ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να τροποποιήσει τη συνθήκη έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα, ότι θα μπορούμε να τα διαβάσουμε, αυτό θα μας βοηθήσει να είμαστε πλήρη μέλη της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μικολάση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Προέρχομαι από τη Σλοβακία. Είμαι γιατρός και ταυτόχρονα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεκριμένα. που έχει στις αρμοδιότητές της και τα θέματα της δημόσιας υγείας. Και έτσι παρακολουθώ όλες τις, προσπάθειες και υποστηρίζω φυσικά όλες τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτών. Υποστηρίζω κάθε προσπάθεια για την ε, κατάργηση των φραγμών ή εμποδίων που βρίσκουν ε, στην καθημερινή του ζωή τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Είναι απαράδεκτη αυτή η φραγμή και τα εμπόδια αποτελούν προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οποιουσδήποτε έχει κάποια μορφή αναπηρίας είναι απαράδεκτο να χρειάζεται να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους εμπόδια στην καθημερινή του ζωή. Και έτσι προσπαθώ και εγώ με την ε, οδηγία για τη βελτίωση των συνθήκων ε, ταξιδίου, είτε πρόκειται για αεροπλάνο, για τρένο, για λεωφορείο, ε, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία συγκεκριμένα, να ε, βοηθήσω κι εγώ από πλευρά μου για τη βελτίωση αυτών των συνθήκων. Πρέπει να εγκριθεί οδηγία, φυσικά στη συνέχεια να εφαρμοστεί και στην καθημερινή ζωή. Επίσης για την αγορά εργασίας μπορούμε να πούμε με το ίντερνετ, ε, με την δουλειά εξ αποστάσεως, με την εργασία εξ αποστάσεως, ε, μπορεί ο εργοδότης μερικές φορές να μην έχει καν συνείδηση του γεγονότος ότι ο εργαζόμενος ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του εξ από το σπίτι του και που έχει μια πολύ καλή κατάρτιση είναι άτομο με, με, με αναπηρία. Γιατί υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα της ε, εργασίας από το σπίτι. Αυτό είναι μια μορφή κατάργησης των εμποδίων και των φραγμών στην καθημερινή ζωή των ΑΜΕΑ. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω ότι είμαι εδώ περισσότερο για να ακούσω τι έχετε εσείς να πείτε, αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πάνω απ' όλα ότι έχετε στο πρόσωπό μας συμμάχους, είμαστε όλοι εδώ και αναζητούμε μαζί σας έναν κοινό παρονομαστή, ένα κοινό πεδίο, ανεξαρτήτως των πολιτικών ή ε, κομματικών ταυτοτήτων μας. Είμαστε εδώ για να σταθούμε στο πλευρό σας. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω ότι οι εκπρόσωποι μας είναι πιο πειθαρχημένοι από τους ευρωβουλευτές. Επόμενος ομιλητής, επόμενη ομιλήτρια είναι μια κυρία από την Ισπανία. Όχι κυρία, Χωσέ Μαρία Σάντσες. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη για την τρόπο που προφέρω το όνομα από το ΣΕΡΜΠΕΙ, το Εθνικό Συμβούλιο για Άτομα με τη της Ισπανίας. Έχετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Στην Ισπανία έχουμε κάποια προβλήματα με την ε, σύμβαση. Είναι θέμα νομικό πρέπει να υπάρξουν τροποποίησεις και το Ισπανικό κράτος να κάνει τις τροποποίησεις που χρειάζεται για να μπορέσει να εφαρμοστεί, να τροποποιηθεί ο ποινικό, για παράδειγμα, κώδικας. Και αλλά εγώ δεν είμαι δικηγόρος, αλλά αυτή η νομική πτυχή είναι περίπλοκη. Και είναι και κάτι επικίνδυνο, γιατί σημαίνει ότι τα άτομα εφόσον κάποια στιγμή ε, κάνουν κάποια παράβαση, κάποιο πλημέλημα κτλ. Ε, δεν μπορούν να έχουν ε, ποινή κάτω από αυτήν που προβλέπεται. Τώρα το κατά πόσο είναι επικίνδυνο ή όχι αυτό πρέπει να το δούμε. Εγώ νομίζω ότι τελικά στρέφεται η κατάσταση σε χρόνια πίσω. Γιατί αντί να βοηθάμε στην ένταξη των αναπήρων, αντίθετα δημιουργούμε παραπάνω προβλήματα Μια τέτοια αντιμετώπιση δεν συνάδει με τη σύμβαση. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι όταν επικυρωθεί η σύμβαση από τα κράτη-μέλη πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή νομική για να μην καταλήγουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι συμβαίνει σήμερα στην Ισπανία με την προσπάθεια εφαρμογής της σύμβασης στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όντω όπως είπε και ο κύριος Κατάνη, διαπιστώνω και εγώ ότι οι εκπρόσωποι μα είναι πιο πειθαρχημένοι από τους ευρωβουλευτές. Ελπίζω και οι ευρωβουλευτές να πειθαρχήσουν στον χρόνο που τους έχουμε δώσει. Χιμένες τώρα από το ΕΛΚ. Παρακαλώ, για δύο λεπτά η κυρία Χιμένες έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που μπορώ να συμμετέχω σήμερα εδώ σε αυτό το φόρουμ. Και θέλω να προσθέσω και εγώ τη δικιά μου τη φωνή σε όλους τους άλλους που μίλησαν για τα βασικά δικαιώματα. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζω όλους όσοι ήρθαν από την Ισπανία. Και υπενθυμίζω ότι το ΣΕΡΜΙΚ, το σχετικό κίνημα της Ισπανίας, κάνει μεγάλη δουλειά. Εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη Δικαιοσύνης και ε, στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Εκεί λοιπόν το θέμα της αναπηρίας με απασχολεί πολύ σε σχέση μάλιστα με τη δικαιοσύνη. Και τελευταία κάναμε μια οδηγία για την προστασία των θυμάτων και έχουμε συμπεριλάβει και ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στις αναπηρίες και στις ειδικέ ανάγκες των θυμάτων που είναι και άτομα με αναπηρίες. Προβλέπονται λοιπόν διάφορα δικαιώματα στην οδηγία αυτή, η ισότητα, η διευκόλυνση στην πρόσβαση και στις ε, δικαστικές διαδικασίες και στην ενημέρωση. Και ιδιαίτερα λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα και δυσκολία κατανόησης και επικοινωνίας που μπορεί να οφείλονται δεχομένω σε κάποιες αναπηρίες, είτε είναι μειωμένη η όραση ή η ακοή. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το άτομο με αναπηρία που είναι και θύμα να μην ε, έχει και παράγωγους λόγους να νιώθει ε, σε αδύναμη κατάσταση. Δηλαδή, μερικές φορές τα άτομα με αναπηρίες που είναι και θύματα εγκληματικής πράξης... είναι δύο φορές θύματα. Πρέπει να έχουν λοιπόν εύκολα πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ιδιαίτερη σημασία δίνουμε και στο θέμα των γυναικών και των ελλείψεων που υπάρχουν στη δικαιοσύνη για την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν πάρα πολλές φορές οι γυναίκες με αναπηρίες είναι ακόμα πιο πολύ θύματα από ό,τι υπόλοιπε. Είμαι στη διάθεσή σας όχι μόνο σήμερα που συζητάμε για τις αναπηρίες, αλλά να ξέρετε και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας είμαι στη διάθεσή σας για συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου μας ζήτησαν το εξή. Προκειμένου να έχουμε την εικόνα στην οθόνη την εικόνα του ομιλητή, όταν φωνάζουμε το όνομά σας, τουλάχιστον εσείς οι εκπρόσωποι, σηκώστε το χέρι σας ε, παρακαλώ για να βλέπουμε που είσαστε. Τώρα έχουμε εκπρόσωπο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Ζωής ε, εν ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρίες. Τζον, παρακαλώ έχετε το λόγο. Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή όπως βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια αδελφοί μας με αναπηρία βρίσκονται σε φυλακή είναι φυλακισμένοι σε ιδρύματα κρατούμενοι σε ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη δεν είναι ελεύθεροι όπως εμείς να συμμετέχουν σε ό,τι δραστηριότητες θέλουν. Δεν μπορούν καν να επιλέξουν τι θα φορέσουν, τι θα φάνε, τι θα πιούν. Και όταν κάθε πρωί που σηκώνονται και κάθε βράδυ που πηγαίνουν στο κρεβάτι, κάποιος ελέγχει τη ζωή τους. Έχουν αγνοηθεί, έχουν παραμεληθεί παρά το άρθρο 19 της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπει ότι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι με αναπηρία και να ζουν αυτόνομα, ελεύθεροι από ιδρύματα, να έχουν την επιλογή του πού θα ζουν, ποιος θα τους στηρίζει, να ζουν εντός της κοινωνίας. Αυτή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πολύ περισσότερο λόγω των σημερινών μέτρων λιτότητας που υιοθετούν πολλές χώρες λόγω των οποίων μειώνονται χρηματοδοτήσεις για την αυτόνομη διαβίωση και άλλες κοινωτικές υπηρεσίες. Αυτό αποτελεί κατάφορη παραβίαση τη ε, συνθήκη για τα άτομα με αναπηρία των ΗΠΑ. Κάνουμε έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να αντιμετωπίσουν αμέσω τα ζητήματα αυτά και να κάνουν έκκληση στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσουν υπεύθυνα τη σύμβαση αυτή των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη βελτίωση των δικαιωμάτων αυτών των ατόμων με αναπηρία και να προστατέψουν τα δικαιώματά μας, να ελευθερώσουν τους αδερφούς μας τώρα. Thank you very much for this very important contribution. Ευχαριστούμε για την πολύ σημαντική σας συμβολή. Είναι πολύ σημαντικό για μας που έχουμε τόσους πολλούς ευρωβουλευτές εδώ. Θα ζητήσω τώρα από την κυρία Μαρία Ιρουγκογιάννη να πάρει το λόγο, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Maria is showing Η Μαρία σηκώνει το χέρι της για την κάμερα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε όλες και όλοι. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας. Και πρώτα απ' όλα μια σκέψη μου, ένα προβληματισμό που θέλω να σας μεταφέρω. Την Κυριακή που μας πέρασε συμμετείχα στη Μαδρίτη στην διαδήλωση του ΣΕΡΜΗ για να καταγγελθεί κάθε αδυναμία που υπάρχει όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην ε, προσαρμογή της νομοθεσίας. Πάρα πολλά άτομα με αναπηρίες στη Μαδρίτη πήγανε με κάθε δυσκολία που όπως καταλαβαίνετε έχουν τα άτομα αυτά για να μετακινηθούν. Και αυτό για να επιμείνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Οι διάφορες δικήσεις έχουν ε, δισταγμούς για τα χρήματα, για τις οικονομίες. Αλλά όπως λέει και το Θέρμη πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι κάτι παραπάνω από απλώς και μόνο προσοχή στην αναπηρία. Η νομοθεσία που ενέκρινε η λευτική Κυβέρνηση το 2007 αναγνωρίζει τη δέσμευση της ε, κεντρικής διοίκησης αλλά και των αυτόνομων κυβερνήσεων να στηρίζουν τα άτομα με αναπηρίε, το περισσότερο από τα οποία είναι γυναίκε. Τα στοιχεία που έχουμε τώρα λένε ότι έχουμε 170.000 και άτομα τα οποία συνεισφέρουν στην κοινωνική ασφάλιση. Τα υπόλοιπα 430.000 μέσω άλλων τρόπων συνεισφέρουν ή επειδή είναι συνταξιοδοτούμενα άτομα. Πάρα πολλοί όμως ε, ε, συγγενείς ατόμων με αναπηρίες που τους προσέχουν δεν έχουν καμία απολύτως εξασφάλιση, κανένα απολύτως έσοδο και καμία απολύτως προστασία. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας αυτό και να προσφέρουμε αξιοπρέπεια στα άτομα αυτά με αναπηρίες στους συγγενείς τους. Το θέμα της εξάρτησης βέβαια έχει άμεση σχέση με την αναπηρία. Πάρα πολλά άτομα ε, που εξαρτώνται από άλλους είναι βέβαια άτομα ανάπηρα, 80.000 στην Ευρώπη, στην Ισπανία επίσης πάρα πολλά, 1.270.000 ε, διαθέτουν ένα πιστοποιητικό αναπηρίας. Και τελειώνω. Είναι αναγκαίο να υπάρξει δέσμευση από τις κυβερνήσεις για ένα ευρωπαϊκό κονδύλι προκειμένου μέσα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια να βοηθώνται τα άτομα με αναπηρίες και να μπορούν να έχουν βοήθεια για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να αναγνωρίζονται τα δικαιώματά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής. Αυστρία. Από το Αυστριακό Εθνικό Συμβούλιο. Η κυρία Ελένη Γιάμαρ. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σας να δούμε πού είσαστε και έχετε το λόγο. Uh, Θα ήθελα να τοποθετηθώ στο θέμα των ε, αναπηριών εν γέννη και ιδιαίτερα των επαγγελμάτων τον Γιατί υπάρχουν πολλά, πολλές σταδιοδρομίες, ιδιαίτερα με πανεπιστημιακές σπουδές, οι οποίες δεν έχουν καν πρόσβαση τα ΑΜΕΑ. Ε, παραδείγματι, η σύμβαση του ΟΙΕ εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ισότιμη δυνατότητα για εξάσκηση επαγγέλματο. Αλλά οι παιδαγωγικέ σχολέ, οι παιδαγωγικέ σχολέ στην Αυστρία δεν εξασφαλίζουν πρόσβαση για τα ΑΜΕΑ. Ή Διαφορετικά μπορεί κανείς να σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία, μεν, χωρίς όμως να μπορεί να πάρει το δίπλωμά του, παρά μόνο ένα πιστοποιητικό το οποίο δεν επιτρέπει να διδάξει σε σχολείο. Σε άλλους τομείς, στα, ε, στα νομικά επαγγέλματα, μπορεί κανείς να πάει να σπουδάσει στη νομική, στις νομικές σχολές και να ολοκληρώσει τις σπουδές του, αλλά δεν είναι σε θέση να ασκήσει επάγγελμα. Ε, του νομικού, του δικηγόρου κτλ. Αυτό ιδιαίτερα αφορά είτε άτομα με τύφλωση είτε άτομα με ε, προβλήματα κοφαλαλίας. Ε, πρόσφατα μάλιστα εγώ είχα προσκαλέσει δικαστές τυφλούς από τη Γερμανία στο Υπουργείο μας, αντίστοιχα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Αυστρία, για να τους δείξω με ε, απτά παραδείγματα ότι είναι δυνατό να είναι κανείς και δικαστής και τυφλός, αλλά αυτό δεν τους έπεισε στο Υπουργείο. Μου είπαν ότι δεν είναι τόσο εύκολο να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Ε, αυτό δεν που με απασχολεί ιδιαίτερω ε, είναι το γεγονός ότι όντως σε ορισμένα κράτη καθίσταται δυνατό το να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του δικαστή κτλ. ακόμα και αν έχει αναπηρία, ενώ κάποια άλλα κράτη το αποκλείουν αυτό σαν δυνατότητα στον τομέα επίσης των ιατρικών επιστημών, αλλά όπως είπα και των νομικών και των παιδαγωγικών, είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η απουσία, αυτή η φραγμή στην πρόσβαση στο επάγγελμα. Τα άτομα με αμαία ξέρουν πολύ καλά ποια είναι τα εμπόδια στο δρόμο τους, τι μπορούν να κάνουν, τι δεν μπορούν να κάνουν και δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουμε άλλα εμπόδια από την νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ πάνω απ' όλα που τηρήσατε το χρόνο σας με ιδιαίτερη ε, πειθαρχία. Θα παρακαλώ την κυρία Ρώστα Εστρέρας να λάβει το λόγο. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα και μάλιστα λίγες μέρες μετά από την ε, μέρα για τις αναπηρίες που είχαμε τη Δευτέρα καλό είναι να δώσουμε τα χέρια και να προχωρήσουμε μαζί για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα για πολιτικές. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ενωθούμε και να προχωρήσουμε υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να ενταχθούν ακόμα καλύτερα στις κοινωνίες μας. Είμαι ευρωβουλευτής. Συμμετέχω στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ανάπτυξη ε, την περιφερειακή ανάπτυξη και θα ήθελα το θέμα αυτό να γίνει προτεραιότητα παντού. Να ενισχυθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, να εφαρμοστεί πλήρως η σύμβαση και η μη διάκριση να αποτελέσει μια εγκάρση αρχή, οριζόντια αρχή που να ισχύει παντού και πάντα σε όλες τις χώρες και να αποτελεί στοιχείο κλειδί κάθε φορά που ε, δίνονται ευρωπαϊκά κονδύλια για να πηγαίνουν στην απασχόληση, στην υγεία, στην εκπαίδευση και των ατόμων με αναπηρίες, γιατί τα άτομα αυτά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχει η κοινωνία. Κάθε κοινωνία η οποία δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να διευκολύνουμε τα άτομα με αναπηρίες, ότι πρέπει να ε, καταργήσουμε τα εμπόδια. Και αυτό θα γίνει αν εφαρμόσουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλες οι χώρες και η Ισπανία είμαι από το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας, κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες για την κρίση, προκειμένου η κρίση να μην σημαίνει και οπισθοχώρηση όσον αφορά τα δικαιώματα αυτά. Και η Ισπανία την κάνει την προσπάθεια, πολύ σημαντική προσπάθεια, ώστε η κρίση να μην σημαίνει και οπισθοχώρηση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Πρέπει και εμείς να υψώσουμε τη φωνή μας προς πάσα κυβέρνηση για να ισχύσει αυτό και στη συνέχεια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, Ιταλία. Από το Ιταλικό Φόρουμ για τις Αναπηρίες, σε πέρο κρυφό. Για δύο λεπτά έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνθήκη αλλάζει το πολιτιστικό πλαίσιο αναφοράς. Επιτέλους είμαστε ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και ως τέτοιο κομμάτι της κοινωνίας πρέπει να απολαμβάνουμε τις εξελίξεις και τα πλεονεκτήματα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Ακόμα σε πολλές χώρες της Ευρώπης είμαστε οι πρώτοι που απομονωνόμαστε λόγω της κρίσης. Από αυτή την άποψη πρέπει να αλλάξουμε πολιτισμική αντίληψη της δικής μας υποστήριξης. Η συνθήκη λέει ότι τα άτομα με αναπηρία γίνονται έτσι διότι η λειτουργική τους διαφορά συναντά εμπόδια, προσκόμματα και διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ζωής. Είναι λοιπόν ευθύνη της κοινωνίας να παρέμβει ώστε να εξαλείψει τα προβλήματα αυτά όχι μόνο στον τομέα της υγείας αλλά και στον κοινωνικό τομέα. Επιπλέον η πρόληψη της ε, αναπηρίας ε, είναι πλεονέκτημα για την κοινωνία. Το 15% σήμερα, 18% του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει κάποια αναπηρία. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους όλοι οι άνθρωποι θα ζήσουν κάποια στιγμή κάποια αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η κοινωνία θα αποκτήσει αναπηρία εάν δεν παρεύει στις γενικές πολιτικές σε παρεμβάσεις αναπτυξιακές. Εμείς ζητάμε να αποτελεσούμε κομμάτι αυτής της εξέλιξης διότι σήμερα δυστυχώς μας ζητούν να έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις χωρίς να έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Από αυτή την άποψη εμείς υπογραμμίζουμε ότι η εξαιρετική παρουσία αυτού του Κοινοβουλίου δείχνει ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες κινητικότητας και χειραφέτησης. Αυτή η χειραφέτηση κινείται προς τη διαφορετικότητά μας ως ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα και σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη είναι διαφορετικοί. Μόνο εμείς υποφέρουμε από στιγματισμό και αποκλεισμό. Γι' αυτό θέλουμε η κοινωνία να αποκριθεί με διαφορετικό τρόπο στα δικαιώματά μας. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω τώρα τον κύριο Βολκαμνόβακ από το Αυστριακό Εθνικό Συμβουλίο Ατομών με Αναπηρία να λάβει το λόγο για δύο λεπτά. Βοηθήστε μας να σας δούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξότιμε κύριε Πρόεδρε, εξότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αξιότιμοι κύριε και κύριοι, πολλές φορές ακούστηκε, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω και εγώ, ότι χρειάζεται μία πλήρης νομοθεσία κατά των διακρίσεων, μια ισχυρή οδηγία κατά των διακρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες είναι το μέσον το οποίο θα μας εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης για όλα τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω και επίσης θα ήθελα να πω ότι και το 2003 ο κύριος Μίχελ Κρίσπελ ε, που είχε, μιλήσει, είχε έρθει και είχε μιλήσει εδώ ένας βουλευτής, ο Μιχαήλ πρέπει το 2003, δυστυχώς φέτος απεβίωσε και θέλω να θυμίσω τη μνήμη του. Σα ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε εκπρόσωπο της Ουγγαρίας. Κύριος Ντάνιελ Ρέκα, ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία. Ντάνιελ Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ονομάζομαι Έντικο Χόρβατ. Είμαι εδώ ως εκπρόσωπος των ατόμων με δυσκολίες μάθησης και θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στα δικά τους προβλήματα. Συστούμε λοιπόν σήμερα μια διεθνή σύμβαση. Είναι πολύ σημαντικό για όλους αυτούς που εκπροσωπώ εγώ. Στα άρθρα 12 και 19 και θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στην δυνατότητα για λήψη αποφάσεων. Εδώ πολλά πράγματα μένουν να γίνουν και να κοιτάξουμε και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον νόμο. Αυτά που αναφέρονται για την δικαιοπρακτική ικανότητα στο άρθρο 12 αλλά και στο άρθρο 13 αποτελούν φυσικά πρόοδο. Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει τη στρατηγική για την διεύρυνση αυτού του πεδίου και βλέπουμε σημαντική πρόοδο να έχει επιτευχθεί πρέπει να κοιτάξουμε την, ε, τις δυνατότητες για υποστήριξη στις συνθήκες ε, διαβίωσης, αλλά με νέο μάτι και πρέπει να υποστηρίξουμε προγράμματα για υποβοηθούμενη, για υποβοηθούμενη διαβίωση. Αυτό το έχουμε κάνει λοιπόν στη χώρα μου και πρέπει να εξασφαλιστούν περισσότεροι χώροι παροχής, ε, παροχής υποβοηθούμενης διαβίωσης. like to ask Mr. Boris Ευχαριστώ. Σουστάσεβιτς τώρα. Ελπίζω να το είπα σωστά. Από το Σλοβενικό Εθνικό Συμβούλιο για δύο λεπτά. Να τηρήσουμε το χρόνο μας όμως. Μετά θα είναι Ερνιφακύρ από τη Γαλλία να προετοιμαστεί. Συστάσεις λοιπόν. Τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αυτή η οικονομική κρίση αυξάνει βέβαια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και επηρεάζει και τη λειτουργία όλων των οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με κάθε μορφή αναπηρίας. Όλους τους σχετικούς συλλόγους, κινήματα κτλ. τα δυσκολεύει. Η χρηματοδότηση των οργανώσεων αυτών γίνεται πολύ αβέβαιη, ακόμη και για τις βασικές τους δραστηριότητες. Οπότε προτείνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να φροντίσουμε να συγκεντρώνονται κονδύλια που να διασφαλίζουν αν μη τι άλλο τη βασική διαβίωση των οργανώσεων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα μπορούσε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για άτομα με αναπηρίες να κάνει μια σχετική πρόταση. Η πρόταση λοιπόν του Σλοβενικού κινήματος για τα άτομα με αναπηρίες είναι ακριβώς ε, αυτό. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ε, χρηματοδότηση μέσω μιας νέας πράξης για τις οργανώσεις για άτομα με αναπηρίες. Έχουμε δηλαδή μια ειδική οργάνωση για τη συλλογή κονδυλίων, ώστε να μπορούν οι δραστηριότητές μας να χρηματοδοτούνται από εκεί. Μόνο έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες και να συνεχίσουμε να βοηθάμε τα άτομα με αναπηρίες ώστε να ζουν ανεξάρτητα. Πάντως οι σημερινές εξελίξεις όσον αφορά την πολιτική που ακολουθείται έχει σαν αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του σημερινού συστήματος και να μας ε, δυσκολέψει ακόμα περισσότερο όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων υπέρ των ατόμων με αναπηρίες. τελικά θα είναι οι αξιωματούχοι οι οποίοι θα αποφασίζουν ε, για μας και για την χρηματοδότησή μας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την σύμβαση του ΟΗΕ και γι' αυτό ελπίζω πως το ψήφισμα θα εγκριθεί σήμερα και ότι θα επηρεάσει κάπως τις παρετέρω εξελίξεις στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Λέω Πρόεδρος. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Αντρέ Φερτιέ από το Γαλλικό Εθνικό Συμβούλιο και επόμενο ομιλητής θα είναι Ingrid Bowman από την Σουηδική Ομοσπονδία για το με Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, τα πολιτιστικά δικαιώματα που υπενθυμίζονται στο άρθρο 30 της ε, συνθήκης του, των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν κεντρικό διακύβευμα. Πρέπει να βγούμε από την κρίση μέσω της ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης, της ευαισθητοποίησης, της συνείδησης των ανθρώπων για την κοινωνία μας. Όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών δικαιωμάτων, παρατηρούμε προόδους σε κράτη, σε κοινωνίες, σε ενώσεις, αλλά οι επιπτώσεις ε, παραμένουν αρκετά περιορισμένες. Εξάλλου, οι βέλτιστες πρακτικές ε, είναι διάσπαρτες δημιουργούν ελάχιστη ανάπτυξη, εξυγχρονισμό και μετάδοση γνώσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα πολιτιστικά μέσα. Και τελικά εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία δεν είναι αυτόνομοι και παραμένουν αποκλεισμένοι από την πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή. Κατά συνέπεια ζητούμε τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας με εκπροσώπους της Κομισιόν του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κινήματος Ατόμων με Αναπηρία, εμπειρογνωμόνων, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες παρακολούθησης της εφαρμογής της συνθήκης για τα πολιτιστικά δικαιώματα και να προσδιοριστούν οι οδοί που θα πρέπει να ακολουθούν για την εφαρμογή της. Όσον αφορά τις, οδού τις ε, μπορούμε ήδη να σκεφτούμε την έκδοση ενός πρακτικού οδηγού για τους επαγγελματίες του πολιτισμού όσον αφορά την προσβασιμότητα του πολιτισμού, την εκπόνηση ε, ρυθμιστικών πλαισίων ε, για τους πολιτιστικούς χώρους τη βελτίωση των κριτηρίων προσβασιμότητας για την επιλεξιμότητα για δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και κάτι βασικό η διασυνοριακή πολιτιστική πρόσβαση ώστε η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών του πολιτισμού να μπορεί να εκφραστεί πλήρως επίσης η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα του πολιτισμού είναι κάτι απαραίτητο δεν είναι δυνατόν πλέον η πρόσβαση στον πολιτισμό να μην αποτελεί προϋπόθεση προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρίες. Τονίζουμε τις αξίες της μη διάκρισης στο πλαίσιο ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Ingrid Μπορμάν από τη Σουηδική Ομοσπονδία να λάβει το λόγο για δύο λεπτά και μετά τον Τζοβάνι Παντοβάνι από την Ιταλία. Σα redan ευχαριστώ πολύ. Από το 2008 μας απασχολεί το θέμα αυτό. Έχουμε μια έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι εκθέσεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Γιατί παρά τις πολλές φιλοδοξίες που έχουμε στην Σουηδία και παρά την ε, θέσπιση της ε, Διεθνούς Συμβάσεως βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί ίσως προς τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ. Χρειάζεται μεταρρύθμιση λοιπόν. Δίνεται υποστήριξη, δινόταν μάλλον υποστήριξη που τώρα έχει περικοπεί, περικόπτονται επίπεδα διαβίωσης, επιδόματα ε, σχετικά με αναπηρία οι ώρες στήριξης, υποστήριξης ε, στον, ε, με, με τις υπηρεσίες υποστήριξης και πρέπει πλέον να σταματήσουν και οι διακρίσεις και η απουσία προσβασιμότητας. Μπορεί να μην έχουμε, μπορεί να υπάρχει αυτή η σύμβαση, αλλά δεν βλέπουμε πολιτικά αποτελέσματα. Αυτή η πολιτική βούληση ή φιλοδοξία που εκδηλώνεται στη Σουηδία δεν μεταφράζεται σε αυτά αποτελέσματα. Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα υλοποιήσουν την ε, Διεθνή Σύμβαση σε κάθε τομέα αρμοδιότητάς τους. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να αποτελέσει κινητήριο μοχλό η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ε, υποχρεώσει με τον τρόπο αυτόν και τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Όπως είπα, έχουμε μάλλον οπισθοδρόμηση σημειώσει στη Σουηδία και πρέπει να θεσπιστούν όργανα ή επιτροπές εποπτείας της υλοποίησης της Διεθνούς Συμβάσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να παρακολουθούν σε κάθε κράτος μέλος ποια κατάσταση επικρατεί και να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση για να έχουμε αντικειμενική κρίση της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει αυτή η πρόταση να ενσωματωθεί και στα πρακτικά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσω. Παρακαλώ τον Τζοβανί Παδοβάνη να κάνει υπομονή για ένα λεπτό. Διότι ο Ευρωβουλευτή Νικόλο Ρινάλντι που έπρεπε να μιλήσει τελευταίο, αλλά χρειάζεται να μιλήσει. Πρώτα του δίνω λοιπόν το λόγο στον ε, κύριο Νικολό Ρινάλντι και μετά στον Τζοβάνι Παδαβάνη. Κύριε Ρινάλντι, έρχεται το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, παρότι ήμουν διατεθειμένος να περιμένω τη σειρά μου. Κανονικά θα μιλούσα στις 12 και 10, αλλά θα μπορούσα να περιμένω ακόμα λιγάκι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι αντιπρόεδρος ε, της τρίτης ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Συμμαχίας ε, Δημοκρατών και Φιλελευθέρων για την Ευρώπη και θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι εκπληκτική. Εγώ προσωπικά, όπως και άλλοι συνάδελφοι της ομάδας μου, δραστηριοποιούμαστε ιδιαίτερα στο θέμα των αναπηριών. Ωστόσο θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί μια μικρή αλλά σημαντική βελτίωση της ποιότητας σε σχέση με όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται διότι βεβαιώνει μια για πάντα το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να έχουν παρουσία εντός ε, των ευρωπαϊκών θεσμοκαϊκών οργάνων και κυρίως το θεσμικό όργανο που εκλέγεται δημοκρατικά. Σίγουρα αυτό εδώ το κοινοβούλιο ε, εποφελείται από αυτή την πρωτοβουλία. Του κάνει καλό να σας υποδέχεται, να ακούει τη φωνή σας, να σας δίνει χώρο. Διαφορετικά θα βρισκόμασταν σε ένα απομονωμένο κάστρο. Αντιθέτως εδώ είναι ο οίκος για όλους τους πολίτες. Ε, στην πολιτική ζωή της Ευρώπης χρειαζόμαστε ακόμα πολλή δουλειά για να γίνουν οι άνθρωποι με αναπηρίες ε, πλήρεις πολίτες ε, στους δημοκρατικούς θεσμούς των χώρων μας. Εγώ σε μια εκλογική εκστρατεία που συμμετείχα το 2009 για τις ευρωεκλογέ. Ε, είχα κάποια συζήτηση με, έναν, με τον Κάρλο Ροσέτη, έναν συνάδελφο με αναπηρία και θα έλεγα ότι η οργάνωση μιας προεκλογικής εκστρατείας είναι εχθρική προς τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Δεν τηρούνται οι προθεσμοί, οι δεσμεύσει, ε, όλα επιβάλλονται πάρα πολύ γρήγορα το ένα μετά το άλλο. Η ταχύτητα του πολιτικού μηνύματος ε, και όλη της υποδομής ε, δημιουργεί προβλήματα σε έναν υποψήφιο με αναπηρία και αυτή είναι μια από τις προκλήσεις του ευρωπαϊκού πολιτικού κόσμου το να ε, γίνουμε πραγματικά ένας πολιτικός κόσμος χωρίς ε, αποκλεισμούς ε, και για όλα τα άτομα με αναπηρίες με ίση εκπροσώπηση όλων των πολιτών. Με λίγα λόγια τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια εξέλιξη του θέματος της αναπηρίας και της σχέσης μεταξύ της αναπηρίας και της κοινωνίας. Αφήσαμε πίσω μας ε, αιώνες διακρίσεων. Ας μην ξεχνάμε από που ερχόμαστε. Ερχόμαστε από έναν μεσαίωνα όπου η αναπηρία ε, καταπιεζόταν, ήταν ε, θεωρείτο ε, αμάρτημα. Για πολύ καιρό η επιστήμη είχε ασχοληθεί, είχε ξεκινήσει να ασχολείται με τις αναπηρίες ε, θεωρώντας τις κάτι ξεχωριστό ένα γκέτο. Έχουμε και την κληρονομιά τον 20ου ε, αιώνα όσους αναπήρους ε, χάθηκαν στο ολοκαύτωμα τη μεγάλη ντροπή του δυτικού πολιτισμού μετά όμως από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο άρχισαμε να ακολουθούμε μια καλύτερη οδό ζητώ συγγνώμη αλλά έχουμε πρόβλημα χρόνου θα πρέπει να ολοκληρώσετε πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να γινόμαστε και πιο διεκδικητικοί. Και σίγουρα το πράτετε εσείς σήμερα οι προκλήσεις ε, δεν είναι οι προκλήσει αναγνώριση των νομοθετικών μέτρων που σε επίπεδο κρατών μελών ή θεσμικών οργάνων τη Ευρώπη μπορούν να ληφθούν. Αυτό γίνεται. Η πρόκληση είναι κυρίω η πλέον εναρμονισμένη εφαρμογή και στα 27 κράτη-μέλη. Παρατηρούμε διαφορές τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά μεταξύ διαφωνών κρατών μελών. Από την άλλη έχουμε την κρίση η οποία πραγματικά απειλεί και διαβρώνει τα κεκτημένα, τα μέχρι σήμερα κεκτημένα. Σήμερα εμείς αντιπροσωπεύουμε ε, ουσιαστικά ένα χώρο όπου θα πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των αναπήρων από τις περικοπές που γνωρίζουμε στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ε, κάτι που να χρησιμοποιηθεί ως ε, ε, μέσο διάσωσης που θα βοηθήσει στην εξέλιξη του είδους μας το να συμπεριλάβουμε τα άτομα με αναπηρία θα αποτελέσει παράμετρο καταμέτρησης του πολιτισμού και της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή εργασία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, πώς βλέπετε, έχουμε μια σημαντική καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να αναβάλουμε την ε, παρέμβαση του κυρίου Χερμαν Φαν Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ίσως οι ομιλητές να μπορέσουν να έχουν ένα-δύο λεπτά ομιλία, εάν οι διερμηνείς μας κάνουν την παραχώρηση να μείνουν άλλα δέκα λεπτά. Μέχρι τις παρατέταρτο όμως που θα πρέπει να διακόψουμε για να αναπαυθούν και οι διερμηνείς. Εάν λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, παρακαλώ τον κύριο Τζοβάνι Παντοβάνι από το ε, Ιταλικό Φόρουμ Αναπηρίων να λάβει το λόγο και ο κύριος Ντέιλι μετά από την Ιρλανδία. Παρακαλώ, Τζοβάνι. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ήθελα να αναφέρω κάτι όσον αφορά τη διατύπωση άτομα με αναπηρία Άκουσα να μιλάμε στη γλώσσα μου για άτομα με διαφορετικέ ικανότητες στα Ιταλικά κατά την ομιλία ενό από του εκπροσώπους τη χώρα μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήθελα να πω ότι αυτή η ορολογία είναι μια ορολογία που δεν μας αντιπροσωπεύει, δεν ορίζει την πραγματική κατάσταση των ατόμων που ζουν με αναπηρίες. Πιστεύω ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι σημαντική η διεθνώ αναγνωρισμένη ορολογία των ατόμων με αναπηρία, όταν μιλάμε γενικά με αναπηρία, πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα γίνεται στη Συνθήκη των ΗΠΑ Εθνών. Όσον αφορά τη σημερινή ημέρα και τη συνθήκη ειδικότερα, ήθελα να σας υπενθυμίσω το άρθρο 27 για την απασχόληση σε σχέση με το τρίτο σημείο της πρώτης ψηφίσματος που θα υιοθετηθεί σήμερα και που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία θα διασφαλίζονται και μέσω των αναθεωρήσεων των εσωτερικών πρακτικών των ευρωπαϊκών θεσμών και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να προβλέπεται η απαραίτητη προσαρμογή για τα άτομα με αναπηρία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτέλεσε το πρώτο θεσμικό όργανο που οργάνωσε εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με αναπηρία. Παρήχε συμβάσει εργασία ε, ε, το πολύ τριών ετών ε, σε άτομα με αναπηρία που επελέγησαν αλλά παρότι ενάρετη αυτή η οδός διεκόπη. Αυτό που ζητώ εγώ είναι δύναμη του άρθρου 27 της συνθήκης όπου προβλέπεται σαφώς ότι κυρίως οι δημοσίοι οργανισμοί θα πρέπει να ε, προβαίνουν σε θετικές δράσεις για να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία. Τι θέλω να κάνει αυτό το κοινοβούλιο, ο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των πολιτών θα ήθελα να εφαρμόσει μια πιο επιθετική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία στο εσωτερικό του, διότι αυτή η ανάγκη γίνεται πιο ορατή εντός ε, των θεσμικών οργάνων, όχι μόνο λόγω της αναπηρίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι έχουν ικανότητες και δεν πρέπει να αποκλείονται από ε, ε δυνάμει των δικαιωμάτων που έχουν ως άτομα με αναπηρία. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής μας από την Ιρλανδία, ο κύριος Νταν Bailey. Κύριε Νταν Bailey έχετε το λόγο. Θα ήθελα σαφώς να επιβεβαιώσω ότι όλα τα μέτρα σήμερα υπονομεύονται καθημερινά και ίσως τα επιδόματα, τα κρατικά επιδόματα, η υποστήριξη από το κράτος μπορεί να μην στηρίζονται σε νομοθετικά μέτρα, να θεωρούνται δεδομένα σε μία χρονική περίοδο, αλλά ε, να μην υπάρχει η κατάλληλη να μην υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες πλαισίου. Και ως εκ τούτου με τις πρώτες περικοπές επηρεάζονται αυτά πρώτα τα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία. Και επηρεάζεται η καθημερινή του ζωή. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε ώστε η κυβέρνηση της Ιρλανδίας να στηρίξει τις, ε, ε, τα επιδόματά μας, να κυρώσει την Διεθνή Σύμβαση και πάνω απ' όλα να νομοθετήσει ώστε να ε, αναγνωριστεί η δικαιοπρακτική ικανότητα για όλους τους πολίτες. Και θα πρέπει να πιεστεί η Ιρλανδική κυβέρνηση ώστε να προχωρήσει το χύτερο δυνατό σε αυτές τις αναθεωρήσεις νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία από την Ουγγαρία έχετε το λόγο. Και μετά ο κύριος Χανσούνγκερ από την Αυστρία. Άικο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Η, Ουγγρα... η Ουγγαρία πριν από μερικά χρόνια υιοθέτησε, κύρωσε καλύτερα την Διεθνή Σύμβαση. Ξεκίνησε όμως πρώτα με την αποδιάρθρωση των μεγάλων θεσμών. Εγώ ε, ιδιαίτερα ασχολούμαι με τα θέματα του αυτισμού και των οικογενειών με αυτιστικά παιδιά. Και θα ήθελα να πω ότι τα άτομα με αναπηρία και οι, οργάνωση, οι οργανώσεις τους μόνο περιορισμένη πρόσβαση στη διαδικασία αυτή την νομοθετική μπορούν να έχουν. Το όχι για μας χωρίς εμάς βλέπουμε να μην έχει αποτέλεσμα ακόμη, να μην εφαρμόζεται. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή της κατοικίας να διεκδικήσουμε. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε να υποχρεώνονται 30-50 άνθρωποι να μένουν μαζί στον ίδιο χώρο, στον ίδια κατοικία και δεν αποτελεί φυσικά αυτό δικαίωμα αναγνωρισμένο από την ε, σύμβαση. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος, ε, ζητώ συγγνώμη, λυπούμε πολύ αλλά αλλά μας υποχρεώνουν οι κανόνες ε, λειτουργίας ε, του Κοινοβουλίου να διακόψουμε το πρωινό μας ε, τώρα, αφού ακούσουμε βέβαια πρώτα τον έναν εκπρόσωπο, το τελευταίο εκπρόσωπο για το πρωινό. Οι υπόλοιποι θα μιλήσουν το απόγευμα, χωρίς όμως να μπορώ να εγγυηθώ ότι θα έχουν όλοι το χρόνο για να τοποθετηθούν. Και βέβαια ευχαριστώ τους ε, διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, που μας έδωσαν ε, περιθώριο χρονικό. Ο κύριος Γκρός έχει το λόγο τώρα από την Αυστρία. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφερθώ στην Ευρώπη του σήμερον και να πω ότι αν αναλογιστούμε ότι το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ε, είναι αφιερωμένο στα διαρθρωτικά ταμεία και ότι πρέπει να οικοδομήσουμε ποτέ την Ευρώπη του αύριον, πρέπει να καταργήσουμε κάθε εμπόδιο στην πορεία, στην ζωή των ΑΜΕΑ και να μην επιτρέψουμε να ε, ανεγερθούν άλλα εμπόδια, άλλη φραγμή. Το, δυστυχώς όμως φαίνεται να φτιάχνουμε μάλλον την Ευρώπη του χτες και όχι το αύριο. Τα μέσα του διαχρονικού του κοινωνικού ταμείου βλέπουμε ότι περισσότερο αφορούν ε, την ε, ε, εξέβρεση θέσεων εργασία για τους ευτυχέστερους πολίτες και όχι τα άτομα με αναπηρίες. Δεν υπάρχει δικημέρινα λοιπόν για τα αμαία στην Ευρώπη. Στις ε, διάφορες επιτροπές και συμβούλια έχουμε μόνο περιθωριακό ρόλο η παρουσία και δεν έρχονται, δεν λαμβάνονται αποφάσεις που να προσφέρουν πόρους οικονομικούς σε άτομα με αναπηρία. Εμείς είμαστε πάντα εκτός. Μόνο εκείνοι που δεν έχουν αναπηρία υποφελούνται αυτών των ευνοϊκών αποφάσεων. Θα ήθελα επίσης ε, να πω ότι τα κονδύλια που προσφέρονται θα πρέπει χωρίς φραγμούς να ε, χορηγούνται στις ενώσεις των ΑΜΕΑ, στις ε, οργανώσεις μας, ώστε να μην έχουμε δυσκολία ως προς την πρόσβαση στα κονδύλια, αυτά και να μπορούμε να τα αξιοποιούμε. Ε, αυτή τη ευχαριστώ θερμά για την παρουσία εδώ. 80 εκατομμύρια με 80 ε, εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες έχουμε στην Ευρώπη και έχουν και αυτά φωνή, έχουν και αυτά λόγο και δικαιώματα. Σας ευχαριστώ θερμά, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος του, της, του πρωινού ε, της πρωινής συζήτησης. Θα πάμε για το μεσημεριανό μας που θα σερβιριστεί στην αίθουσα Γεχούντι Μενουχίν. Σας καλώ να επιστρέψετε στις 2 και 20. Δύο και είκοσι ακριβώς για να συνεχίσουμε και να καλύψουμε το χαμένο χρόνο.